Uh, Εάν είσαστε έτοιμοι ως ΛΥΜΠΕ, γιατί ξέρω ότι μερικοί από εσά πρέπει να διευθετήσουν θέματα ταξιδιού κλπ. Θα ήθελα να σας κάνω ορισμένες ανακοινώσεις πριν περάσουμε στην ψηφοφορία της έκθεσης Μακοβέη. Παρακαλώ όσοι θέλουν να αποχωρήσουν να το κάνουν. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι ως προς το 2.1, το 2.1 έχει προστεθεί στην ημερήσια διάταξη σε σχέση με ελέγχους ε, για τις τράπεζες δεδομένων στα εξωτερικά σύνορα. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, τροποποιείται η ημερήσια διάταξη. Ε, ως πως, ε, όπως πως γνωρίζετε, τα κροατικά, μαλτέζικα και γαλλικιακά δεν είναι διαθέσιμα σήμερα. Ως προς τις κατεξουδότηση πράξεις έχουμε λάβει τρεις δυνάμει του κανονισμού 98-2013 σε σχέση με την εμπορία των πρόδρομων ουσιών. Αν θεωρείτε λοιπόν ότι μπορείτε να το δεχτείτε, θα υποβάλουμε μία ε, πρόταση ψηφοφορίας. 7 Δεκεμβρίου είναι η ε, προθεσμία και εάν αντιδράτε και δεν δέχεστε τις κατεξιοδότηση πράξεις θα πρέπει να το αναφέρετε μέχρι τότε. Ε, έχουμε τη, τις εξής κατεξιδότηση πράξης ε, κανονισμός της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό 98 κάθετος 2013 σε σχέση με την σκόνη αλουμινίου στις πρόδρομες ουσίες και ο κανονισμός πάλι που αντικαθιστά το 98 2013 σε σχέση με την ε, ε, σκόνη μαγνησίου και, ε, και μαγνησίου και εξάειδρου μαγνησίου στον κατάλογο των πρόδρομων ουσιών. Υπάρχει λοιπόν και η πρόταση που τροποποιεί στην, ε, τον 562 του 2006 σε σχέση με τις ε, βάσεις δεδομένων στα εξωτερικά σύνορα. Θέλετε κυρία Μακοβέη να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία διανύσαμε και δύσκολες στιγμές, καθώς και καλές, και στο τέλος φτάσαμε σε μία εξισορροπημένη λύση που αποδεχτήκαμε όλοι. Ελπίζω αυτός ο κανονισμός να μας οδηγήσει σε μια ασφαλέστερη Ευρώπη και Ευρώπη, μια Ευρώπη όπου διασφαλίζονται οι ελευθερίες. Ευχαριστούμε. Άρα ψηφίζουμε τώρα επί του κειμένου το οποίο συμφωνήθηκε ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 45 ψήφισαν υπέρ και 8 κατά. Καμία αποχή. Να συγχαρούμε την κυρία Μακοβέη. So, colleagues, that's the end of voting Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες προς το παρόν συνάδελφοι και τώρα προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. Εάν δεν σας απασχολεί σας παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχως. Σημεία 3 και 4 της ημερήσιας διάταξης σε σχέση με το σύστημα εισόδου-εξόδου για την καταχώρηση δεδομένων ως προς τις, ε, τα ευφυή e σύνορα, το πακέτο αυτό έχει μία προθεσμία. Παρακαλώ να αποχωρήσετε. Όσοι δεν όσους δεν απασχολεί αυτό το θέμα. Σε 6 Απριλίου η Επιτροπή ενέκρινε την ε, νέα νομοθετική πρόταση, την αναθεωρημένη και ε, έναν κανονισμό σε σχέση με ένα σύστημα εισόδου-εξόδου. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Ντίας Τεμέρα, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για τις δύο εκθέσεις. Κύριε Ντίας Τεμέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω δύο σχέδια έκθεσης σε σχέση με το πακέτο εφιών συνόρων σε σχέση με τη θέσπιση συστήματος εισόδου-εξόδου στο χώρο Σέγγεν και θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε 142 τροπολογίες για την επόμενη έκθεση για την αλλαγή του συστήματος ε, εισόδου-εξόδου. Έχουμε 17 τροπολογίες συνολικά. Όπως γνωρίζετε και οι δύο ε, εκθέσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και γι' αυτό οι τροπολογίες ε, και των δύο εκθέσεων έχουν, ε, έχουν επίπτωση και στις δύο. Οι μεγάλες ε, ροές προς την Ευρώπη δείχνουν την ανεπάρκεια του συστήματος ελέγχου στα εξωτερικά μας σύνορα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να επιδράσει και τις αλλαγές που θα επέλθουν τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε το σύστημα διαχείρισης εισόδου-εξόδου για να είναι πιο αποτελεσματικό αλλά και πιο ασφαλές. Εάν δεν κάνουμε κάτι μεσοπρόθεσμα θα καταρρεύσουν τα σημεία εισόδου-εξόδου και γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν πολλές επενδύσεις σε υποδομή και προσωπικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ροές αυτές. Η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος εισόδου-εξόδου θα ευεργετήσει τους επιβάτες στα σύνορα και παράλληλα θα μπορούν να εξυπηρετηθούν, δηλαδή οι επιβάτες, ε, καλή την πίστη, για να φτάσουμε σε μία συσσωρόπηση, μεταξύ διευκόλυνσης και ασφάλειας. Αλλά επίσης ε, θα ευεργετήσει τους υπεύθυνους ε, υποδομών και θα αυξήσει τη συνδεσιμότητα με άμεσα οικονομικά και έμεσα οικονομικά ευεργετήματα. Θέλουμε λοιπόν να βελτιστοποιήσουμε τα σημεία εξόδου-εισόδου και αυτό αφορά και τους μεταφορείς, το δίκτυο μεταφορών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα στοιχεία που ενυπάρχουν στο σύστημα. Όπως βλέπετε και στην έκθεσή μου, προσπαθώ να ε, καθησυχάσω τις ανησυχίες που υπάρχουν, γιατί θέλουμε να εξασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων. Τα δύο σχέδια έκθεσης αφορούν το εξής του στόχου τις υποδομές, την διαλειτουργικότητα τα βιομετρικά στοιχεία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την περίοδο διατήρησης των δεδομένων και τις επιπτώσεις τους επιβάτες και τους μεταφορείς, καθώς και το όλο σύστημα διαχείρισης. Η στόχη μου ήταν η εξής, να γίνει πιο εύρωστο το σύστημα νομικής ασφάλειας, και νομικού ελέγχου σε σχέση με τα σημεία και τον χρονισμό στις εισόδους-εξόδους και έχω επιβάλει και τροπολογίες έτσι ώστε ο Ευρωπαίος Επόπτης Προσωπικών Δεδομένων να ενισχυθεί στη δράση του και να νιώθουν ασφαλείς οι επιβάτες. Για παράδειγμα, θα ζητούμε δακτυλικά αποτυπώματα μόνο υπάρχει, όταν υπάρχει θέμα ασφάλειας. Επίσης, να ενισχύσουμε τα σώματα ασφάλειας έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση εξ αρχής στο όλο εγχείρημα τηρώντας ε, τις προδιαγραφές νομικής ασφάλειας, έτσι ώστε να συμμετέχουν μόνο εκείνοι τους οποίους ε, αφορά το σύστημα. Προσπαθήσαμε να ευθυγραμμίσουμε αυτό το κομμάτι με τον ε, κανονισμό της Europol και την ασφάλεια δεδομένων, καθώς και το ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη προσωπικών δεδομένων, του κ. Μπουταρέλη. Θα ήθελα επίσης να υπάρχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας έτσι ώστε να υπάρχει προσβασιμότητα υπό συγκεκριμένους όρους και σε περίπτωση που θα υπάρχουν τεχνικές ελλείψεις. Επίσης θέλω να ευθυγραμμίσουμε το σύστημα εισόδου-εξόδου με το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων και άλλα σχέδια νομοθετικού περιεχομένου που σχετίζονται με μελλοντικές ε, ε, διαβουλεύσεις όπως το Eurodac και το ETIAS. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να ευθυγραμμίσουμε άρθρα και ορισμούς. Θα προσπαθήσω να έχουμε ε, διεθνή πρότυπα σε σχέση με τα δακτυλικά αποτυπώματα έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται κατά 100% για τους στόχους που προορίζονται και για να μην έχουμε επικαλύψεις και για την συλλογή και αρχιοθέτηση των δεδομένων. Θα συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα ε, στα πλαίσια εκθέσεων για τις ε, διάφορες φάσεις του συστήματος. Η Εουλίσσα είναι ε, το πλαίσιο πραγμάτωσης και υλοποίησης του συστήματος. Η ΕΟΛΙΣΑ είναι ένας ειδικό οργανισμός, ο οποίος ε, φέρει ευθύνη μέσα στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του κύκλου του συστήματος. Θα ήθελα το σύστημα εισόδου-εξόδου να ισχύσει το 2020, να είναι λειτουργικό. Γι' αυτό θα πρέπει να εργαστούμε πολύ στενά κατά το πρώτο εξάμεινο του επόμενου χρόνου. Αυτό όχι μόνο για το μέλλον του συστήματος, αλλά και για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει σε άλλα συστήματα, όπως το σύστημα πληροφοριών έφιας. Για τις τροπολογίες προτείνω προθεσμία τη 10η Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Επειδή όμως μεσολαβούν και τα Χριστούγεννα, και μου το ζήτησαν και συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας προτείνω να παρατείνουμε λίγο την προθεσμία μέχρι την Πέμπτη στις 2 το απόγευμα, έτσι ώστε στις 20 Φεβρουαρίου να το ε, εξετάσουμε το όλο θέμα και την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου να ψηφίσουμε και μέχρι πρώτη, την 1η Μαρτίου υπό Μαλτέζικη Προεδρία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις για τη συνεργασία τους ήταν απόλυτα απαραίτητη. Ευχαριστώ. Thank Σε ευχαριστούμε πολύ που αναγνωρίζετε και το έργο των σκιωδών και ξεκινούμε τους σκιώδεις παρακαλώ εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Αγουστίν Δεμέρα Σίτη για αυτή την έκθεση, για την εξαιρετική συνεργασία μέχρι σήμερα. Καταρχήν κάποιες πρώτες γενικού χαρακτήρα παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Από την αρχική πρόταση ήταν μακρά η πορεία επισκεφθήκαμε διάφορους μεθοριακούς σταθμούς, κάναμε μια πιλωτική μελέτη και τώρα υποβάλλεται μια νέα πρόταση ενώπιόν μας. Το πρόγραμμα αυτό δεν προβλέπεται για συχνούς ταξιδιώτες, για ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά και είναι κρίμα θεωρώ εγώ αυτό. Πρόκειται για τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα, καλό αυτό γιατί μειώνονται τα κόστη, από την άλλη όμως πλευρά η πρόταση σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής ε, παρεκκλίνει και μια μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης των στοιχείων προβλέπεται και τα λοιπά. Πρέπει να πω ότι ο κύριος στόχος αυτής της πρότασης είναι η διαχείριση των συνόρων, των διασυνοριακών διελεύσεων και η διευκόλυνση όσον αφορά τους ταξιδιώτες και να δούμε ποια είναι η διάρκεια και ποια είναι η παράβαση όσον αφορά εκείνους που ε, παρατείνουν τη διάρκεια της ε, διαμονής τους ε, ανεφάδιας, overstayers. Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας τίθεται στο ίδιο σημείο εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά πρέπει να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση. Όλοι οι διασυνοριακά ταξιδεύοντες θεωρούνται ως μια, σε μια κατηγορία και θεωρούνται πολύ ύποπτοι και σύμφωνα με τις νέες διατάξεις έκθεση Μακοβέη την οποία μόλις ψηφίσαμε το ίδιο θα ισχύει και για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η καταπολέμηση της εγκληματικότητας δεν μπορεί να επηρεάζει τη διέλευση συνόρων από ταξιδιώτες. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό σε σχέση με τη δουλειά μας. Δεν έχω πιστεί για αυτά τα θέματα. Δεν μπορούν να πείθουν τα επιχειρήματα των κρατών και μάλιστα να, έχει πρόσβαση, να έχουν πρόσβαση ιδιοκτικές αρχές σε όλα αυτά τα στοιχεία συλλήβδιν. Πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση μεταξύ νόμιμων ταξιδιωτών που τηρούν τις ε, διατάξεις της νομοθεσίας και νόμιμα μεταβαίνουν από μια χώρα στην άλλη και μάλιστα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα να διαφοροποιούμε μεταξύ αυτών και των άλλων που είναι overstayers και παραβιάζουν τη διάρκεια αυτή. Πρέπει να δούμε λοιπόν κατά πόσον, για ποια διάρκεια θα αποθηκεύονται τα στοιχεία αυτά. Και άσχετα ποια μορφή θα πάρει το τελικό κείμενο, το σύστημα διαχείρισης, FES σύστημα διαχείρισης συνόρων, Smart, Border System, θα πρέπει να μας κάνει να μπορούμε να είμαστε, να διαφοροποιούμεθα έναντι της προσέγγισης ε, των θεμάτων ταξιδιωτών. Θα πρέπει περισσότερες πληροφορίες να δίνονται στους ταξιδιώτες, να γίνει αυτή η προσπάθεια από πλευράς μας για τα ταξίδια αυτά και τους όρους. Ε, πρέπει να γνωρίζουν το τι ισχύει, να γνωρίζουν τις διατάξεις και πρέπει επίσης και να μπορούν να τηρούν και να μην παραβιάζουν αυτό το κανονιστικό πλαίσιο. Πρέπει να βρούμε ένα ευφυές αποτελεσματικό τρόπο προσέγγισης όλων αυτών των θεμάτων. Οι νέες διατάξεις θα μπορούσαν φυσικά να οδηγήσουν στο να επιδεινωθεί η κατάσταση, ιδιαίτερα σε κάποιους εκτεθειμένους ε, μεθοριακούς σταθμούς. Στην ε, Σλοβενία, για παράδειγμα, υπάρχει πληθώρα συρροή δηλαδή τέτοιων ταξιδιωτών σε κάποιους ε, σταθμούς θα πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά τα οποία πράγματι είναι σημαντικά. Ευχαριστώ. Thank ε, ευχαριστούμε για την ως ο Σκιώδης από πλευράς τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ΙΣΙΑ υποστηρίζει και πάντα υποστήριζε το σύστημα εξόδων, εισόδων-εξόδων θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί πριν από την κατάργηση των, ε, στα εσωτερικά σύνορα στην Ένωση. Αλλά έστω, τέλος καλό όλα καλά, κάλιο αργά παρά ποτέ. Η ευφυής διαχείριση συνόρων για αυτούς που συχνά ταξιδεύουν και ένας καλύτερος έλεγχος των εξωτερικών συνόρων μας είναι αναγκαίες προϋποθέσεις. Οι αρχές επιβολής του νόμου, οι αρχές της τάξης πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία για να είναι αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρήσιμα και η περίοδος αποθήκευσης αυτών των στοιχείων πρέπει να είναι επαρκής ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά από τις αρχές ασφαλείας. Είναι καλά διατυπωμένες οι προτάσεις από πλευράς του εισηγητή του κυρίου Δίας Δεμέρα. Κάτι λιγότερο θα μας εξέπλητε φυσικά. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα το ότι ο κύριος Δίας Δεμέρα έκανε προσπάθεια να συγχρονίσει να θέσει σε, παράλληλο, σε παράλληλη τροχιά αυτό τον κανονισμό σε σχέση με τα όσα ισχύουν από πλευράς Eurodac για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδους κανονισμοί και κανόνες να εναρμονίζονται μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης και εναρμονισμού. Είναι πολύ ενθαρρυντικό και προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία με τον εισηγητή και του σκιώδη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Και από πλευρά σας, Άλντε, παρακαλώ, σκιώδης εισηγήτρια, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολλή δουλειά που επένδυσε όχι μόνο για αυτό το κείμενο αλλά και για τις συναντήσεις με τους σκιώδεις και με τους ε, ε, πραγματογνώμονες. Ευχαριστούμε θερμά. Σε σχέση με το σχέδιο έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να γίνεται σαφές ότι κάνουμε λόγο για υπηκόους τρίτων χωρών. Ωστόσο κάποια προβληματικά θέματα τα οποία αφορούν την πρόταση της Επιτροπής, αφορούν την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεν επιλύονται επαρκώς. Η νέα πρόταση όσον αφορά την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά για τις αρχές ασφάλειας προβλέπει μια δυσανάλογη περίοδο αποθήκευσης η οποία ισχύει στο σύνολο του εύρους αυτής της πρότασης και δίνει μη επαρκή ε, πρόσβαση σε σχέση με μηχανισμούς προστασίας δεδομένων. Η προηγούμενη πρόταση είχε ένα θέμα υπόψη, την διαχείριση συνόρων σε σχέση με τους ελέγχους ε, όσον αφορά αυτούς τους ταξιδιώτες. Διαρωτώμεθα πώς μπορούμε με τόσο πολύμορφο πλαίσιο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. Η πρόταση όσον αφορά πρώτον που έχουμε καταθέσει αφορά τον περιορισμό του εύρους ε, και την θέση εντάξει και δεύτερον να ισχύουν μόνο αυτά τα οποία αναλογικά είναι απόλυτα αναγκαία και τρίτον να περιοριστεί η περίοδος αποθήκευσης δεδομένων. Προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία με τον εισηγητή και τους άλλους σκιώδεις και ελπίζω ότι στο τέλος θα βρεθεί μια σωστή ισορροπημένη συμβαστική λύση. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Άλμπερτ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εισηγητή για το έργο που επετέλεσε σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Επίσης για την δυνατότητα όπως ζητήθηκε να υπάρξει κάποιος χρόνος για τις τροπολογίες περισσότερος όλοι ευχαριστούμε για αυτό δεύτερον αυτό που ήταν αφαγιών ανέφερε και άλλος συνάδελφος για την περίοδο αποθήκευσης θα ήθελα να το αναφέρω και εγώ για τις δυνατότητες οι διοκτικές αρχές, οι αρχές ασφάλειας να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα για άλλες χρήσεις, για άλλους σκοπούς. Και στα δύο αυτά θέματα έχουμε εναλλακτικέ λύσεις που εκπονούνται για αυτή την πρόταση που είναι πιο αναλογικές για τους στόχους αυτού του χαρτοφυλακίου. Και στο τέλος τέλος είναι πιθανόν ότι διαφορετικά αν δεν ακολουθήσουμε αυτές τις προτάσεις θα υπάρξει η δημιουργία μιας ευρύτατης τεράστιας τράπεζας δεδομένων με μεγάλη περίοδο αποθήκευσης πράγμα το οποίο δεν θα ήταν αποτελεσματικό για τη λειτουργία, για τους στόχους που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε εμείς με αυτή τη ε, δυνατότητα και θα ήταν και πολύ πιο δαπανηρό σε σχέση με ένα άλλο εναλλακτικό σύστημα όπως προτείνεται και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η περίοδος όσον αφορά την ε, ε, διάρκεια αποθήκευσης ε, δεν νομίζουμε ότι είναι η πιο εύθετη. Θα πρέπει να δούμε αυτό που είπε η Τάνια Φαγιόν και σε αυτό να παραμείνουμε διαφοροποίηση δηλαδή εκείνων που ταξιδεύουν νόμιμα και σε τακτή βάση και εκείνους τους άλλους που ε, ίσως δεν τηρούν αυτά τα ε, δεδομένα. Είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό. Και τέλος αλλά εξίσου σημαντικό πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι αυτό το σύστημα ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές, θα ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές προστασίας δεδομένων όπως ε, ε, τα συναφή που έχουμε συζητήσει για την προστασία δεδομένων μέχρι σήμερα. Η προστασία δεδομένων στα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ζητήσαμε να ακολουθείτε και ζητάμε και οι επιχειρήσεις να το σέβονται πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ευχαριστώ. Άλλο συνάδελφος θέλει να παρέμβει και έτσι Μπορούμε να επανέλθουμε στον κύριο Ντίαστε Μέρα τώρα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Απλά δύο λόγια να πω που εντάσσονται στο πλαίσιο της αναγκαίας ευγένειας και να, των ευχαριστειών. Για την Τάνια Φαγιών θα ήθελα να πω ότι δεν μπορώ να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπε. Γνωρίζει πολύ καλύτερα και πολύ καλά αυτό το χαρτοφυλάκιο και έτσι Χωρίς ε, καμιά αμφιβολία σίγουρα χρειάζομαι την υποστήριξή σου Τάνια Φαγιόν και χρειάζομαι επίσης και τα ερωτήματα και αμφιβολίες που διατυπώνεις από πλευρά σου για να προχωρήσουμε σε σχέση με Γιούση και έχει και από πλευράς ε, των παρατηρήσεων πολύ μεγάλη πείρα για το χαρτοφυλάκιο. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τα λόγια σου και νομίζω ότι καλώς βαίνουν οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για να συγχρονιστούν τα συστήματα εισόδων-εξόδων με τα άλλα συστήματα όπως Eurodac για παράδειγμα. Θα ληφθεί λοιπόν υπόψη αυτό στην Αγγελική Αγγέλικα που είναι καινούρια σε σχέση με αυτό το χαρτοφυλάκιο αλλά είναι πολύ, με πολύ ενεργό τρόπο συμμετέχει. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις που έκανε. Θα έχουμε ευκαιρία να τις συζητήσουμε Κάνει αναφορά η Αγγέλικα στην, δυσανάλογη, στην μη ανάλογη σχέση που μπορεί να υπάρχει για την περίοδο αποθήκευσης των ε, δεδομένων. Είναι κάτι το οποίο είναι ε, αντικείμενο κοινό αυτό ως παρατήρηση. Θα αποτελέσει αντικείμενο εξειδικευμένης και σε βάθος συζήτησης και εξέτασης. Την ανησυχεί την Αγγελική και εμένα επίσης η σωστή προσπελασιμότητα πρόσβαση των δυνάμεων ασφαλείας, ε, των αρχών ασφαλείας σε ένα τέτοιο σύστημα. Όπως όμως και με το προηγούμενο σύστημα αυτό δεν είναι ένα υπουσιώδες δευτερεύον θέμα. Είναι ένα θέμα που μπορεί να συγκριθεί με το υπόλοιπο της νομοθετικής πρότασης. Και Ζαν που είναι αρχή και πράγματι ε, έχει κύρος για αυτά τα θέματα στην Ευρωβουλή και πρόκειται για στρατευμένο άτομο για τα θέματα αυτά Βοηθά πολύ λοιπόν αυτή η στάση και μου άρεσε αυτό που είπες ότι αυτό το νομοθετικό, αυτή η νομοθετική δέσμη μέτρων πρέπει να σέβεται την ε, αναλογικότητα στο, στην αντιμετώπιση των προσωπικών δεδομένων. Στη σωστή κατεύθυνση λοιπόν στοχεύουμε έτσι. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς πορείας και ευελπιστώ ότι θα είναι γόνιμη για όλους. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστούμε κύριε Διαθεμέρα. Θα έλεγα ότι έχουμε την ευλογία να έχουμε ένα καλό εισηγητή και σκιώδης εισηγητέ για να γίνεται έτσι καλή δουλειά και αυτό είναι προνόμιο και προτέρημα. Και έτσι ως αφετηρία μπορούμε να συνεχίσουμε με θετικό τρόπο. 12 Ιανουαρίου η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Και γνωρίζετε ότι θα υπάρξουν πολλές τροπολογίες που θα κατατεθούν κύριε Ντιεύτε μέρα. Ευχαριστώ για αυτή την καλή εκκίνηση. Ευχαριστώ και εσάς και τους Κιώδης. Ευχαριστώ συνάδελφοι. So, colleagues, again, um, we go to... Συνάδελφοι, και πάλι πάμε στον Διαθεμέρα, πάλι στον κύριο Διαθεμέρα, για το πώς έχουν οι διαπραγματεύσεις του τριμερούς διαλόγου <clears throat> και πώς εξελίχθηκαν όσον αφορά υπηκός τρίτων χωρών και το θέμα θεωρήσεων, διαβατηρίων για την ε, διέλευση συνόρων και το τι ισχύει όσον αφορά αυτά τα θέματα. Και εισαγωγικά, εχθές να πω ότι στις 7 Δεκεμβρίου όσον αφορά τους ε, ε, τριμερείς διαλόγους που έλαβαν χώρα και Ζητώ από τον κύριο Ντίας Μέρα να μας ενημερώσει λοιπόν σχετικά με τα τεκτενόμενα. Παρακαλώ. Πολύ καλά, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Λοιπόν, με ικανοποίηση και χαίρομαι ότι μπορώ να πληροφορήσω τα μέλη της Επιτροπής μας για το θετικό αποτέλεσμα του τελευταίου τριμερούς διαλόγου. Το πρώτο που θα ήθελα να αναφέρω είναι να ευχαριστήσω να ευχαριστήσω τις διάφορες πολιτικές ομάδες της Ευρωβουλής και σε αυτό το κεφάλαιο θα ήθελα να αναφερθώ σε όλους αλλά ξεχωριστά στην Πριζίτ κυρία Τσίμπελ που όπως έχουν τα πράγματα με την πολιτική της ομάδα και η ίδια και υπήρχαν διαφορές ουσίας όσον αφορά θέματα αυτής της έκθεσης και επιβλήθηκε, επικράτησε στο τέλος θα έλεγα το ευρωπαϊκό πνεύμα που την εμπνέει και τη διαπνέει όσον αφορά την προσέγγιση για τα ευρωπαϊκά θέματα. Έγιναν παρεμβάσεις που τις εκτιμώ και ευχαριστώ για αυτές και τη σοσιαλιστική, σοσιαλδημοκρατική ομάδα. Το ίδιο πρέπει όμως να πω σε σχέση και με τους φιλελεύθερους, το ίδιο επίσης πρέπει να πω και σε σχέση με την ECR, τους μεταρρυθμιστές, ε, δημοκράτες μεταρρυθμιστές που είχαν μια, μια πολύ δραστήρια συμμετοχή. Εδώ υπήρχαν και οι πράσινοι που είχαν ε, συμμετοχή και ευχαριστώ όλους που βοήθησαν να αποτροχοπεδθεί, να απελευθερωθεί αυτό το θέμα. Ήταν πάρα πολύ σύνθετο και περίπλοκο σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το θέμα. Γιατί, διότι <clears throat> σε σχέση με την επίλυσή του απορρέων τα θέματα για τη Γεωργία και την Ουκρανία στον αφορά την αναθεώρηση καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίων και για την απελευθέρωση αυτών των ε, θεμάτων αυτής της έκθεσης πρέπει να δοθεί ένα σαφές αδιαμφισβήτητο μήνυμα για αυτούς τους λαούς, τους πολίτες αυτών των εθνών και ευχαριστώ λοιπόν όλους για την προσπάθεια και επίσης και τη γραμματεία μας και όλους τους βοηθούς μας και συνεργάτες μας και την ομάδα μας και τις άλλες ομάδες που συμμετείχαν με αποφασιστικό τρόπο. Ε, μέχρι την τελευταία στιγμή διήρκεσε η αγωνία γι' αυτό. Να υπενθυμίσω, υπήρχε μια, ε, ε, ένα θέμα επίμαχο το οποίο ε, κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα χθες σε σχέση και με το Παρίσι και ευτυχώς από το Παρίσι πήραμε την έγκριση το πράσινο φως. Και ευτυχώς αυτό συνεισέφερε στο να αποτροχοπεδηθεί τελεσίδικα το θέμα αυτό. Ήταν κάτι το αναγκαίο αυτό και είναι σημαντικό. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για τον πολύ κομψό τρόπο με τον οποίο μας ενημερώσατε. Πραγματικά πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα από τα πιο ευαίσθητα νομοθετήματα που θα μπορούσε να είχατε ποτέ αναλάβει. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και να ευχαριστούμε και όλους τους συναδέλφους στα πλαίσια της ΛΥΜΠΕ, οι οποίοι όπως είπατε σας βοήθησαν προκειμένου να ευοδοθεί το όλο νομοθέτημα. Δεν είπα βέβαια το πιο προφανές στην αρχή, ότι μπορούμε πλέον να ψηφίσουμε την πράξη αυτήν και αυτό προβλέπεται στα πλαίσια της σημερινής ψηφοφορίας που θα έχουμε με συγκεκριμένο κατάλογο ψηφοφοριών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για το εξαιρετικό σας έργο και για το χρόνο που αφιερώσατε για το νομοθέτημα αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή εκπρόσωπος από τη Σλοβακική Προεδρία που ενδεχομένω να θέλει τώρα να πάρει το λόγο. ενδεχομένω να αξίζει αυτή τη στιγμή να ακούσουμε και την παρέμβαση της Προεδρίας. Εν συντομία παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τα όσα είπατε ότι όντως ε, ο φάκελος αυτός ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος, ε, αντιμετωπίστηκε κατά προτεραιότητα όχι μόνο από το Συμβούλιο, από την Προεδρία του Συμβουλίου δηλαδή, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την Επιτροπή σας για την επιλογή του αξιότατου ε, εισηγητή, ο οποίος έδειξε ότι ήταν έτοιμο να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μια συμβαστική πρόταση, η οποία μα επέτρεψε τελικά να μιλάμε σήμερα για επιτυχία. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και τους χειώδεις εισηγητές, οι οποίοι προφανώς βοήθησαν τον εισηγητή σας και βέβαια να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον επικοδομητικό της ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Να ολοκληρώσω όμω το σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολλά πράγματα θα μπορούσε να θίξει κανείς σχετικά με το φάκελο αυτό. Προ στιγμήν όμω νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσω αυτό το σημείο. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ και εμεί χαιρόμαστε πολύ που ακούμε τα όσα είπατε εκ μέρου τη ε, Προεδρία, το ότι καταφέραμε να πετύχουμε τελικά έναν κοινό στόχο και πάλι προ όλε τι πολιτικέ ομάδε και προ όλου του εργαζόμενου, πολιτικέ ομάδε που ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό. Για άλλη μια φορά απευθύνω τι ευχαριστίε μου, καθότι ε, ο φάκελο αυτό ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο και δύσκολο. Δεν ξέρω αν ο κύριο Διά Ντεμέρα θέλει να προσθέσει κάτι ακόμα. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Για να ολοκληρώσουμε πρόεδρε, επίσης και εγώ θέλω να υπογραμμίσω, να τονίσω τη δουλειά και τον επαγγελματικό χαρακτήρα με το οποίο εργάστηκε η Σλοβακική Προεδρία. Ήταν δύσκολη, δυσχερής διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, μέσα σε ένα πλαίσιο κατανόησης και επαγγελματική θετικής αντιμετώπισης ε, ε, ε, εκτιλήχθηκε. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνώρισε πώς έπρεπε να διατηρήσει τις αρμοδιότητες της, γνώριζε η Επιτροπή πώς έπρεπε να φερθεί επαγγελματικά, διασφαλίζοντας τον θεσμικό χαρακτήρα και την διαθεσμική συνεργασία. Ευχαριστώ και το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντίας Δεμέρα και απευθύνω και εγώ τις ευχαριστίες μου ω πρόεδρο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 6 της ημερήσια διάταξης, Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εδώ είχα υποβάλει ένα αίτημα η δική μα Επιτροπή προκειμένου ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να εκπονήσει δύο μελέτες, δύο γνωμοδοτήσεις όσον αφορά πρώτον την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κέντρα υποδοχή και ταυτοποίηση hot spots τη Ιταλία και τη Ελλάδο. Η δεύτερη δε γνωμοδότηση έχει να κάνει με την επίπτωση που θα μπορούσε να έχει για τα παιδιά ο νέος κανονισμός για το Δουβλίνο. Ας ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Νέσπορ, ο οποίο θα μα παρουσιάσει την πρώτη γνωμοδότηση για τα Hotspot και συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μολνάρο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την δεύτερη γνωμοδότηση που έχει να κάνει με το νέο σύστημα του Δουβλίνου. Στη συνέχεια, αγαπητά μέλη, θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε και εσεί παρατηρήσεις όσον αφορά τι δύο αυτέ γνωμοδοτήσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα προβληθούν, θα προβληθούν και κάποιες διαφάνειες στα πλαίσια της παρουσίας του κύριου Νέσπορ. Περιμένουμε λίγο λοιπόν μέχρι να τακτοποιήσουμε τεχνικά ζητήματα σχετικά με τις διαφάνειες αυτές. Μιλήσουμε λοιπόν για τα hotspots. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι έτοιμη και η παρουσίαση με τις διαφάνειες. Ας ακούσουμε λοιπόν την παρουσίαση της πρώτης γνωμοδότησης από τον κύριο Νέσπορ όσον αφορά τα hot spots στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στην Ιταλία και την Ελλάδα. Κύριε Νέσπορ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας παρουσιάσω στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ την πρόσφατη αυτή γνωμοδότησή μας, δύο μάλιστα γνωμοδοτήσεις που μας ζήτησε η Επιτροπή σα, Εγώ θα σας παρουσιάσω την πρώτη γνωμοδότηση που έχει να κάνει με την κατάσταση των μορδών δικαιωμάτων στα hot spots της Ιταλίας και της Ελλάδας. Και ο συναδελφό μου κύριο Στάμα Μολνάρ θα κάνει τη δεύτερη παρουσίαση όσον αφορά τη γνωμοδότηση για την προτινόμενη αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, επικεντρώμενο, επικεντρώμενος περισσότερο επιπτώσεις που μπορεί να έχει στους ασυνόδευτού ανήλικου και στα παιδιά. Δεν θα επιμείνω στο τι είναι hotspot και πώς λειτουργεί, γιατί νομίζω ότι γνωρίζετε ήδη πολύ καλά. Σας συνάντησα ορισμένου στην Λέσβο τον Ιούνιο, όπου μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία δική σας ήρθε για να επισκεφθεί το hotspot που βρίσκεται εκεί. Ξέρω λοιπόν ότι γνωρίζετε όλοι πολύ καλά τα βασικά χαρακτηριστικά και τη βασική δομή των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, εγώ θα ήθελα εν συντομία να πω ορισμένα πράγματα όσον αφορά τη γενικότερη φιλοσοφία της γνωμοδότησης αυτής Ποια είναι η προσέγγιση όσον αφορά τα hotspots. Στόχος εδώ πέρα είναι να έχουμε μια συντονισμένη δράση, μια συντονισμένη ανταπόκριση όσον αφορά τη μαζική έλευση προσφύγων μέσω θαλάσσης στην Ιταλία και την Ελλάδα. Και η προσέγγιση αυτή είναι διτή. Από τη μία πλευρά έχουμε ένα συντονισμό της δράσης όσον αφορά τις διαδικασίες εκείνες που θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να ομαδοποιηθούν σε έναν χώρο. Αναφέρομαι εδώ πέρα στην καταχώρηση των ε, μεταναστών, των προσφύγων και την λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να ευθυγραμμίσουμε όλες τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν και να δούμε επίσης ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί, αν θα είναι κατάσταση, αν θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία επιστροφής και το καθεξής. Προσπαθούμε επίσης να οματοποιήσουμε λίγο τη δράση των παραγόντων επιτόπου. Είδαμε ότι υπάρχουν έχουν μια πολύ μεγάλη παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ΕΑΖΟ και από την Frontex, αλλά και από την Europol. Και η γνωμοδότηση βέβαια καταγράφει το γεγονός αυτό. Λέμε ότι όλες αυτές οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες εξακολουθούν και έχουν ένα ρόλο υποστηρικτικό, προσπαθώντα να βοηθήσουν τις εθνικές δημόσιες αρχές. Παράλληλα όμως οι δράσεις τους έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο σε κάποιου τομείς όπως για παράδειγμα η διεκπαιρέωση των αιτήσεων ε, διεθνούς προστασίας και ασύλου. Θεωρούμε λοιπόν ότι ε, στην πράξη υπάρχει μια κοινή ευθύνη μεταξύ ευρωπαϊκών αρχών και εθνικών αρχών όσον αφορά τις λειτουργίες των hotspots. Υπάρχουν κάποια κενά όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που μπορεί να μην έχουν να κάνουν άμεσα με τη λειτουργία των ε, Ευρωπαίων παραγόντων. Παρόλα αυτά συμβάλλουν κατά της νομιμότητας της δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης η ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν από την αρχή παρών επιτόπου στα hot spots αυτά, παράλληλα με εθνικές αρχές, προκειμένου να παρακολουθήσει την προστασία, την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μια συγκεκριμένη εμπειρία και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Μια ακόμα γενική παρατήρηση, η γνωμοδότηση, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας όσον αφορά τα hot spots, τόσο όσον αφορά τη γενική κατάσταση, όσον αφορά τη φύση των μεταναστευτικών ροών, αλλά και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο έχουν επηρεαστεί τα hot spot από άλλες εξελίξεις. Και εδώ πέρα βέβαια έχουμε να κάνουμε και την ε, δήλωση και τη συμφωνία του Μαρτίου 2016 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουρκίας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα ελληνικά hot spot έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στις λειτουργίες επιστροφής, επαναπατρισμού ορισμένων προσφύγων προς την Τουρκία. Και βέβαια και οι αιτήσει ε, ασύλου καταχωρούνται, καταγράφονται, άμεσα στα hot spots στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στα hot spots της Ιταλίας. Η γνωμοδότηση λοιπόν εξετάζει τα hot spots ως ένα πιλωτικό τελικά πρόγραμμα, ως ένα πρόγραμμα άντλησης διδαγμάτων, γνωρίζοντας ότι οι πρακτικές που ακολουθούνται αυτή τη στιγμή δεν προβλέπονταν εξ αρχής όταν ε, άρχισαν να λειτουργούν τα hot spot. Έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις από τότε που στήθηκαν τα hot spot αυτά. Παρ' όλα αυτά λέμε ότι υπάρχουν σημαντικά κενά όσον αφορά την προστασία και την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και βλέπετε εδώ πέρα στις διαφάνειες κάποια από τα κενά αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει. Το πρώτο σημαντικό θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι το ζήτημα της πρόσβασης στο καθεστώς διεθνούς προστασίας. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στο καθεστώς αυτό. Αυτό είναι άλλωστε και ένας από τους πρωταρχικούς στόχους των hotspot. Πάρα πολλά άτομα τα οποία φτάνουν τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα ουσιαστικά ζητάνε άμεσα διεθνή προστασία. Κάνουν άμεσα αίτηση για άσυλο. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα όλες τις διαδικασίες καταχώρησης, καταγραφής, διεκπαιρέωσης των αιτήσεων ασύλου και εδώ πέρα θεωρούμε ότι τα hot spots συμβάλλουν θετικά. Παράλληλα όμως και ιδίως στην Ελλάδα και εδώ αναφέρομαι σύν από τα κέρια σημεία της γνωμοδότησης τα hotspot εκεί έχουν συμφοριστεί κατά κάποιο τρόπο όσον αφορά το ζήτημα της διεκπαιρέωσης των αιτήσεων ασύλου ακριβώς επειδή υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις όσον αφορά τις ισορρευμένες αυτές αιτήσει. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις στην καταχώρηση των αιτήσεων αυτών, που σε ένα βαθμό βέβαια το φαινόμενο αυτό βελτιώθηκε, χάρη και στην εργασία της ΕΑΖΟ και του προσωπικού της. Βλέπουμε όμως ότι το ζήτημα αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό εξαιτία της ιεράρχης προτεραιοτήτων ως προς την εθνικότητα των προσφύγων. Ξέρουμε ότι οι Σύριοι ήταν αυτοί οι οποίοι κατά προτεραιότητα γινόντουσαν δεκτοί όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων εσύλου. Μετά όμω τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Τουρκία δόθηκε προτεραιότητα στην επιστροφή προσφύγων προ την Τουρκία και ακολουθούν στη συνέχεια κάποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών από χώρε οι οποίε δεν αποτελούν προτεραιότητα, όπω για παράδειγμα οι προερχόμενοι από το Πακιστάν. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν και κάποιε ε, άλλε εθνικότητε που δεν αποτελούν προτεραιότητα, οι υπήκοοι των οποίων περιμένουν πολλέ φορέ ακόμα και έξι μήνες στα hot spot, ουσιαστικά από τότε που υπεγράφει η συμφωνία με την Τουρκία. Περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί στα hot spot χωρίς να έχει διεκπαιδευτεί καμία αίτησή του. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολλέ αρνητικέ επιπτώσει. συμφόρηση των ε, hot spot αυτών, αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τα παιδιά και ιδίω όσον αφορά του ασυνόδευτου ανηλίκους, και υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τη δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν καταγραφεί πλήρω όλα τα άτομα τα οποία αιτούνται άσυλο. Τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν και προβλήματα στι προσπάθειέ του να επανορθούν με τι οικογένειέ του. Και κάτι ακόμα εξίσου σοβαρό είναι ότι ε, το ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί πλέον άνθρωποι που περιμένουν στα hot spot αυτά οδηγεί πολλές φορές σε τεταμένες καταστάσεις, ακόμα, ακόμα επίσης και σε βία φαινόμενα, σε εκδήλωση βίας μεταξύ των ε, διαμενόντων στα hot spot αυτά. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να αποσυμφορήσουμε κατά προτεραιότητα τα hot spot. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των παιδιών τα οποία διαμένουν στα hot spot, εδώ πέρα έχουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην γνωμοδότησή μας. Χρησιμοποιούμε και κάποια στατιστικά δεδομένα. 37% των αφήξεων του 2016 στην Ελλάδα είναι παιδιά ουσιαστικά. Αντιστοιχούν σε παιδιά. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε παιδιά τα οποία φτάνουν με τις οικογένειές τους, αλλά και σε παιδιά τα οποία φτάνουν ε, ασυνόδευτα ή και σε παιδιά τα οποία φτάνουν χωρίς τους γονείς τους, αλλά συνοδευόμενα από άλλους ενήλικες. Η κατάσταση λοιπόν των παιδιών αποτελεί και στα δύο hot spot και στις δύο περιπτώσεις hot spot Ιταλίας και Ελλάδας βασική μας προτεραιότητα. Θα έλεγα ότι το πιο καυτό ζήτημα είναι τα μη συνοδευόμενα παιδιά. Κάποια στατιστικά δεδομένα τους πρώτου 9 μήνες του 2016 περίπου 19.000 ασυνόδευτα παιδιά φτάσανε στην Ιταλία. Και στην Ελλάδα όμως και στην Ιταλία τα ασυνόδευτα παιδιά, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία πρέπει να πηγαίνουν σε ειδικέ δομέ μετά την άφηξή του, προκειμένου να προστατευτεί το μίσον συμφέρον του παιδιού και γενικότερη ευημερία των παιδιών, πράγμα το οποίο όμω δεν συμβαίνει πολλέ φορέ. Δηλαδή, ακριβώ επειδή δεν υπάρχουν αυτέ οι εξειδικευμένε δομέ ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ιταλία. Στην Ελλάδα τα αριθμητικά δεδομένα μας δείχνουν ότι μόνο το, το ίμιση των παιδιών στους καταλόγους αναμονής καταφέρουν να περάσουν σε ειδικευμένες δομές. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά παραμένουν στα hot spot, μαζί με τους ενήλικες δηλαδή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια σειρά προκλήσεων. Μένοντας τα παιδιά στα hot spot, ουσιαστικά βρίσκονται υπό το καθεστώς προσωρινών μέτρων κυδαιμονίας ακριβώς επειδή δεν έχουν τους γονείς τους ή τους επίσημους κυδαιμόνες τους. Ουσιαστικά είναι αρμόδιοι δημόσιοι υπάλληλοι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν προσωρινά την κυδαιμονία των παιδιών. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ πέρα συγκεκριμένου ε, ε, ε, εισαγγελείς ε, εξειδικευμένου σε ζητήματα παιδιών στην Ελλάδα ή ανθρώπου που προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, Δημάρχου, για παράδειγμα στην Ιταλία. Οι άνθρωποι αυτοί σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικευμένοι σε ζητήματα επιμέλεια παιδιών και δεν μπορούν να αναλάβουν πλήρω το καθήκον αυτό τη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού. Όταν για παράδειγμα ένας δήμαρχος από μια συγκεκριμένη πόλη πέρα από τα καθήκοντά του θα πρέπει να αναλάβει και την επιμέλεια και δαιμονία για 200 παιδιά, καταλαβαίνετε ότι το εγχείρημα αυτό καθίσταται πάρα πάρα πολύ δύσκολο και προφανώς ο άνθρωπος αυτός δεν θα καταφέρει εξατομικευμένα να βοηθήσει τα παιδιά αυτά. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει είναι το ζήτημα της, του υψηλού βαθμού προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών Ζήτημα το οποίο απαιτείται προκειμένου τα παιδιά αυτά να μην αποτελέσουν σε καμία περίπτωση αντικείμενο κακομεταχείρισης. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε ποιες λύσεις έχουν βρεθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Έχουμε εδώ πέρα ένα σύστημα κυδαιμονίας. Ουσιαστικά τα παιδιά κρατούνται στα hot spot αυτά, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από τα hot spot στις περισσότερες περιπτώσεις. Και βέβαια εδώ πέρα δεν ισχύουν οι κατάλληλες συνθήκε. Τα παιδιά δεν θα έπρεπε να ζουν για παραταμένο χρονικό διάστημα στα hot spot. Δεν υπάρχουν, όπω είπαμε, απαραίτητε υποδομέ υποδοχή, Δεν προβλέπεται συγκεκριμένα συστήματα επίσημη τυπική εκπαίδευση και τίθενται και κάποια ζητήματα ασφάλεια. Ακούσαμε για περιπτώσει βιασμού ασυνόδευτων παιδιών σε ορισμένα hot spot και δεν υπάρχει επίσης και εξειδικευμένο προσωπικό για την προστασία των παιδιών στα hot spot. Μολονότι λοιπόν υπάρχουν κάποιε βελτιώσει που έχουν λάβει η χώρα και προβλέπονται βελτιώσει τόσο από τι ελληνικέ όσο και από τι ταλικέ αρχέ, για παράδειγμα και στι δύο χώρε προβλέπεται μια νομοθετική αναθεώρηση τη εθνική νομοθεσία όσον αφορά το προσωρινό σύστημα κυδαιμονία. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο βελτίωση. Θα πρέπει κατά προτεραιότητα να βελτιώσουμε την κατάσταση των παιδιών, των παιδιών στα hot spots και στις δύο αυτές χώρες. Ας δούμε τώρα και την τελευταία διαφάνεια της παρουσίασής μου. Το τρίτο ζήτημα το οποίο θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε στα πλαίσια της γνωμοδότησης έχει να κάνει με τα δύο φύλλα και την αντιμετώπιση τους. Ακριβώς όπως έχουμε παιδιά στα hot spots, έχουμε και πολλές γυναίκες και καταλαβαίνετε ότι σε πάρα πολλά hot spots υπάρχουν νέοι υγιείς άντρες, όπως πολύ συχνά παρουσιάζονται, και η διαφοροποίηση αυτή δεν λαμβάνεται πάντα υπόψη στα hot spots. Όπως και τα παιδιά έτσι και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ε, πολύ σημαντικούς κινδύνους ενώ ζουν στα hot spots και είχαμε και φαινόμενα βίας, φαινόμενα βίας βάση του φύλου και υπάρχει και οι γυναίκες ανήκουν ουσιαστικά σε ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού πολλές φορές ε, έχουν υποστεί ψυχολογικά τραύματα ακριβώς επειδή μπορεί να έχουν χάσει την οικογένειά τους ε, ενώ ταξίδευαν, ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ιταλία ή στην Ελλάδα Πολλές φορές οι γυναίκες αυτές έχουν πέσει θύμα παράνομης διακίνησης. Έχουμε πάλι στατιστικά δεδομένα από διεθνείς οργανισμούς που μας δείχνουν ότι όχι μόνο οι γυναίκες αυτές έχουν πέσει θύμα παράνομης διακίνησης, αλλά πολλές φορές αποτελούν και αντικείμενο σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικής εμπορίας. Είναι πολύ σημαντικό εδώ πέρα πάλι να χρησιμοποιούνται εξειδικευμένε υπηρεσίε, οι οποίε δυστυχώ απουσιάζουν. Τώρα, ποιε λύσει μπορούμε να βρούμε. Θα ήταν εύκολε κάποιε λύσει. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλέ περισσότερε γυναίκε εργαζόμενε στα hot spots θα μπορούσαν για παράδειγμα να ασχολούνται με τι συνεντεύξει αυτέ, οι οποίε γίνονται για τους περισσότερους πρόσφυγες, για παράδειγμα γυναίκες εργαζόμενες να ασχολούνται με τη συνέντευξη γυναικών προσφύγων, αυτό θα βοηθούσε τις γυναίκες αυτές να ανοιχτούν περισσότερο και να μιλήσουν με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και με μεγαλύτερη άνοιση για κάποια ζητήματα. Θα μπορούσαν κατά αυτόν τον τρόπο να έχουν καλύτερη πρόσβαση στη διεθνή προστασία. Υπάρχουν και κάποια προευαίσθητα ζητήματα όπως η λήψη δακτυλικών αποτυπμάτων που πάλι τα δακτυλικά αποτυπώματα των γυναικών θα ήταν καλύτερο να τα λαμβάνουν γυναίκες εργαζόμενες στα hot spots. τα κάποιες νυχτερινές περιπολίες. Άλλα θέματα περιπολιών κατά τη νύχτα για παράδειγμα ή για τα θέματα προστασίας των θυμάτων για να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι όσον αφορά τα καταλήματα για τη διασφάλιση της προσωπικής ζωής και όσον αφορά τουαλέτες για παράδειγμα που όταν είναι η μία δίπλα στην άλλη και χρησιμοποιούνται και από τα δύο φύλλα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Πολλές γυναίκες ε, στα πως δεν πάνε, σε, δεν θέλουν να καταλήγουν σε αυτές τις ε, τουαλέτες ε, και σε σχέση με τα θέματα λουτρών για παράδειγμα ή συναφών χώρων πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες προσπάθειες ε, και σε σχέση με τη διασφάλιση των στόχων που εκθέτουμε στην γνωμοδότησή μας για να μπορούν να καλυφθούν αυτά τα ζητήματα από τις εθνικές αρχές εν κατακλείδη, συμπαράσματι συμπεράσματι, ενώ μπορούν στο μέλλον τα hot να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο για να αντιμετωπίζονται οι νέες αφήξεις, είναι ιδιαίτερη ανησυχία κάποια θέματα όσον αφορά για παράδειγμα και τα παιδιά που πρέπει επιτακτικά να, να επιληθούν από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο εθνικό επίπεδο. Έχει ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διασφάλιση των προτεραιοτήτων αυτών και που θα είναι σεβαστές όπως πρέπει. Και υπάρχει και υποχρέωση να υποστηρίζονται τα κράτη-μέλη με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ώστε οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούν εκεί να λειτουργούν υπό σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε ένα σωστό περιβάλλον. Επαρκούμε σε αυτά. <clears throat> Ίσως μακρηγόρησα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε και για τον χρόνο. Εμείς συγκεκριμένα ζητήσαμε να παρουσιαστεί αυτή η γνωμοδότηση και είμαστε ευγνώμονες ε, για την ε, ε, παρουσίαση αυτή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν αρκετοί συνάδελφοι και θα παρέμβουν με τη σειρά που ζήτησαν τον λόγο και περνάμε στην πρώτη παρέμβαση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Όσον αφορά τα παιδιά στα spots, παιδί αναφέρεται ως όρος ε, για οποιονδήποτε είναι κάτω από 18 ετών και αν ναι, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες ε, επαλήθευσης και πώς διαφοροποιείται σε σχέση με ένα πραγματικό παιδί πραγματικά δηλαδή ηλικιακού φάσματος παιδικής ηλικίας με έναν άλλον που μπορεί να είναι 17 ετών αναφέρεται ότι 37% όσον αφορά τις αφήξεις 2016 στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει 37% όλων των αφήξεων ε, καλύπτουν αυτή, αυτό το φάσμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας. Είναι πάντα ενδιαφέρον να διαβάζει κανείς τις μελέτες σας, διότι πραγματικά επικεντρώνονται στα ζητήματα και καθώς βρισκόμαστε στο επίκεντρο της διαδικασίας αναθεώρησης του συστήματος ασύλου στην Ευρώπη, Εξαρτόμαστε από την υποστήριξή σας για να πάνε όλα καλά, γιατί την τελευταία φορά δεν τα καταφέραμε και σε σχέση όλας και με την σύμβαση του Δουβλίνου υπήρξε πάγωμα της όσον αφορά συγκεκριμένες χώρες. Όσον αφορά την αύξηση, την κατάσταση των παιδιών είχαμε στο Κοινοβούλιο μια ανταλλαγή απόψεων, μια κρόαση με πολλές ΜΚΟ από την Ιταλία και την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται εκεί και αυτό που αναφέρεται είναι ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί πια διότι θα πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε, διότι τα παιδιά χάνονται καθοδόν. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που δεν ξέρουμε τι απέγιναν στην Ευρώπη και έχουν απολεστεί, σύμφωνα με στοιχεία της Europol. Αν τώρα η κατάσταση είναι όπως αυτή που μας επισημάνθηκε από τις ΜΚΟ που δρούν στην ε, Ιταλία και την Ελλάδα στα χόσπος ότι συλλαμβάνονται παιδιά για, χωρίς καμιά αιτία και κρατούνται, στήθενται υποκράτηση επί μήνες πολλές φορές και κανένας δεν λαμβάνει υπόψη τον ευάλωτο χαρακτήρα των παιδιών αυτών, ιδιαίτερα των ασυνόδευτων παιδιών. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα μπορούσαν να παραμένουν υπό τέτοιε ε, συνθήκες τα παιδιά και να ζουν έτσι και να μην προσπαθούν να δραπετεύσουν και στη συνέχεια ίσως με αυτόν τον τρόπο χάνονται κιόλα. Γι' αυτό δεν γνωρίζουμε τι απογίνονται. Πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πράγματα για να μπορέσουμε να αποθαρρύνουμε να συνεχίσουν να μετακινούνται προς ένα άλλο κράτος μέλος ε, σε μια βάση μη νόμιμη ή που να μην βρίσκεται σε ε, νόμιμα πλαίσια. Και πρέπει όλα αυτά βέβαια να αλλάξουν. Ερώτησή μου, ποια είναι τα δικά σας βιώματα, τι είδατε ότι γίνεται σε σχέση με την ε, κατάσταση ε, κυδαιμονίας αυτών των παιδιών. Είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ ευάλωτα αυτά τα παιδιά και είναι ο αποφασιστικός χαρακτήρας που θα πρέπει αυτός προτεραιότητα να επικρατεί όλα τα άλλα που κάνουμε και πώς διασφαλίζουμε λοιπόν στη συνέχεια ότι ουσιαστικά θα μπορούμε να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων σε σχέση με τις υποχρεώσεις μας έναντι τέτοιων ευάλωτων ε, όντων όπως είναι τα προστάτευτα, συνόδευτα παιδιά. Υπάρχουν και άλλες ευάλωτες ομάδες, αλλά επιλέγω να επικεντρωθώ στην ευάλωτη ομάδα των παιδιών αυτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχετε τώρα εσείς τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά Ακούγεται και είναι απίστευτο ότι συζητάμε επί μήνες ολόκληρος την κατάσταση αυτών των παιδιών που είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αυτό που συμβαίνει. Γιατί αυτό που συμβαίνει με αυτά τα παιδιά εκεί είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Είναι ένα έγκλημα κατά των βασικών αρχών ε, που διέπουν ε, την ανθρωπιστική δράση. Τι εννοούμε τώρα όταν λέμε κατεπηγόντως. Κατεπηγόντως σε μια, δυο μέρες, τρεις, σε μερικές εβδομάδες, σε κάποια χρόνια ή τριάντα χρόνια. Τι εννοούμε εδώ όταν λέμε κατεπηγόντω να γίνει κάτι. Ποιο είναι υπεύθυνο για αυτά τα ανθρωπιστικά εγκλήματα. Ποιο προσήχθη δικαστήριο ποτέ για τέτοια πράγματα. Είναι ένα ζήτημα της Ελλάδα και τη Ιταλία. Όχι. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί εθνικά. Είναι κάτι οικουμενικό, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό. Και σε σχέση με την Προεδρία και όλα, στο αναφέρω, την παρουσία και όλα και της ε, Προεδρίας της Σλοβακίας και η πρωτοβουλία λέει της Βρατισλάβας και με τους κανονισμούς. Τώρα συζητήσατε σε σχέση με το Συμβούλιο τον κατεπήγοντα χαρακτήρα που έχουν αυτά τα πράγματα π.χ. για τα παιδιά και για τις λύσεις. Ποιος μπορεί να παράσχει οι λύσεις. Οι λύσεις δεν μπορούν να βρεθούν και να διοργανωθούν εδώ. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως από μια ομάδα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί για να παρακολουθεί τα θέματα. Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η συνθήκη του Δουβλίνου που θέτει υποχρεώσεις ε, στις χώρες όπως την Ιταλία και την Ελλάδα δεν λειτουργεί, δεν είναι το εύθετο πλαίσιο. Δηλαδή ένας αστυνόμος, αστυνομικός στην Ελλάδα θα είναι υπεύθυνο για την ζωή, για τη μοίρα χιλιάδων παιδιών. Αφάνταστο, ασύλληπτο αυτό με βάση αυτή την ανάλυση τι προτείνετε εσείς για να επιληθεί το πρόβλημα. Έχετε κάποια ιδέα ποια θα ήταν η ιδανική λύση. Πώς θα προβλεπόταν μια τέτοια λύση από πλευρά σας για παράδειγμα. Ευχαριστώ πρόεδρο σας ευχαριστούμε. Πολλοί από μας συμμερίζονται υπό αυτή την έννοια αυτές τις τοποθετήσεις για τις ερωτήσεις που τέθηκαν σε σχέση με όλα αυτά για να δοθεί ίσως να φωτιστεί το θέμα και από πλευράς Βίξτρον που ετέθη πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι ώστε από πλευράς του δυναμικού που υπάρχει όσον αφορά το, τις δράσεις για τους πρόσφυγες υπάρχουν ενδείξεις και τεκμήρια για το τι θα μπορούσε για παράδειγμα να γίνει όσον αφορά και τα υψηλότατα επίπεδα βίας και όσα γίνονται όσον αφορά τους ε, διακινητές ανθρώπων και την κατάσταση στα hot spots. Είναι μια κατάσταση που έχει εξελιχθεί και έχει οξυνθεί σε σχέση με τους πρόσφυγες αυτούς. Και τα όσα αναφέρονται σε σχέση με το εύρος αυτής της κατάστασης η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχουν ενδείξεις ε, τεκμήρια για την, το πόσο ξύνεται η κατάσταση σε σχέση με το ανθρωποεμπόριο και για το πόσο όλα αυτά επηρεάζουν την κατάσταση αυτών των ατόμων και τι συμβαίνει ακριβώς. Ε. Και το άλλο είναι το θέμα της Ευρωπόλ. για την εξέταση ακριβώς αυτών των ε, ε, κατηγοριών ή των όσων έχουν ε, παρουσιαστεί. Κάνει λόγο η Ευρωπόλ για εθνικές αρχές κρατικούς υπαλλήλους που επιλέγονται από την Ευρωπόλ για την δράση για την προστασία παιδιών και την διαμεσολάβησή τους. Πώς εσείς βλέπετε αυτή την κατάσταση Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αναφέρατε όχι μόνο την πρόοδο που επετεύχθη στην Ιταλία και την Ελλάδα, επίσης αναφέρατε και κάποια κενά που υφίστανται και πολύ διαφορετικούς λόγους για τους οποίους βλέπουμε να υφίστανται κενά και χάσματα και δεν θα πρέπει να θεωρείτε ότι αυτά ισχύουν μόνο για την Ιταλία και την Ελλάδα. Κάνουμε λόγο για τα θεμελιώδη δικαιώματα λοιπόν. Θεμελιώδη δικαιώματα για αυτούς τους ανθρώπους στα hot spots, στο, στους χώρους πρώτης άφηξης και για ανήλικους και για άλλες ευάλωτες ομάδες. Ποια είναι η δική σας προοπτική υπό την άποψή σας. Αν αρχίσουμε τώρα να οδηγούμε σε επιστροφές ε, πρόσφυγες που καταλήγουν στη Γερμανία, Γαλλία, αλλού, αλλά πρώτα όμως είχαν ε, αφηθεί, είχαν φτάσει στην Ελλάδα. Πώς το βλέπετε αυτό, αν ξεκινήσουν πολλά κράτη-μέλη να ε, επιστρέφουν αυτά τα άτομα στην Ελλάδα, πώς μπορεί να συνεισφέρει να βελτιωθεί η κατάσταση ή πώς ίσως θα επιδεινωθεί κιόλα η κατάσταση με κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα εις βάρος των παιδιών. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε χρόνο γιατί τελειώσαμε τις εκθέσεις ε, πολύ γρήγορα. Η κυρία Βίκστρομ μπορεί να υποβάλει και άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε για τη γενοδορία σας, κύριε Πρόεδρε. Όταν έχουμε χρόνο γίνεται κάτι τέτοιο. Ξέρετε, σήμερα το πρωί προχωρήσαμε πολύ γρήγορα με όλα τα σημεία. Δεν θα ε, ήθελα να ε, μιλήσω μόνο για τα πεπειραμένα μέλη. Ε, βάση περιπτώσει ανέκυψε και ένα άλλο ζήτημα, η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων που εγκρίθηκε το 2011, όπου έχει εφαρμοστεί και για την Ιταλία και για την Ελλάδα και υπάρχουν ειδικέ διατάξεις για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά και πολλοί από τους ανθρώπους για τους οποίους μιλάμε εμπίπτουν σε αυτή τη κατηγορία. Η ΦΡΑ είδε πως ε, ε, υπάρχει πραγματική εγγύηση τήρησης αυτών των δικαιωμάτων στα hot spot γιατί εγκρίθηκε αυτή η οδηγία και πρέπει να ισχύσει και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για τις ε, ερωτήσεις, εξειδικευμένες ερωτήσεις. Ξέρω ότι ε, δεν έχετε εντολή να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά θα θέλαμε την άποψή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν υπερβάλλω. Αυτό δείχνει ότι παρίστανται τα μέλη που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα, κάτι το οποίο εκτιμούμε ιδιαίτερα. Θα απαντήσω στο μέτρο που μπορώ. Το πρώτο ερώτημα είναι ένα ερώτημα ουσίας, αλλά ίσως και αντίστροφα. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία φτάνουν στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει περιορισμός μετακινήσεων. Ιδιαίτερα ε, ισχύει αυτό για τα παιδιά στα ε, νησιά που αποφασίζουν να μην δηλωθούν ως παιδιά. Γιατί γνωρίζουν ότι με την παρούσα κατάσταση το να είναι κανείς παιδί είναι περιορισμός και όχι ευεργέτημα αν είναι κανείς 17χρονος και ασυνόδευτος που είναι παιδί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα γνωρίζει ότι είναι πολύ καλύτερα να πει ότι είναι 18. Το 37% είναι μία εκτίμηση κατά προσέγγιση με βάση τα δεδομένα των Ηνωμένων Εθνών, της ΥΠΑ της Αρμοστίας δηλαδή μετά τις δηλώσεις ε, κατά την προσέλευση των, ε, στα hot spot. Γίνονται εκτιμήσεις αν κάποιος δηλώσει ότι είναι παιδί και δεν το πιστεύουμε, τότε γίνεται μία επανεκτίμηση, αλλά αυτό το 37% αφορά την κατάσταση πριν από την εκτίμηση, αλλά σίγουρα δεν θα είναι χαμηλότερος ο αριθμός. Ε, σκόπιμο όμως αυτό που αναφέρατε. Τώρα, σε σχέση με αυτά που ρώτησε η κυρία Βίκστρομ, σε σχέση με τα παιδιά. Βέβαια, ε, όλες οι ερωτήσεις αφορούν τα παιδιά. Κάτι το οποίο δείχνει ότι καταλαβαίνετε για, ως προς τη βαρύτητα του ζητήματος. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη στον οργανισμό. Ως προς τα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί, δεν έχω ε, μιλήσει ακόμα επί του θέματος. Το οι 10.000 είναι συντηρητικό, συντηρητική προσέγγιση. Είναι πολύ ψηλότερος δυστυχώς ο αριθμός έμπρακτα πολλές φορές ε, λέγεται ότι κρατούνται χωρίς λόγο τα παιδιά, δεν λαμβάνουμε υπόψη τον ευάλωτο χαρακτήρα τους. Δυστυχώς οι αρχές ε, θεωρούν ότι κρατούν τα παιδιά για την προστασία τους, γιατί δεν έχουν μέσα άλλα μέσα στη διάθεσή τους. Άρα δεν είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται με τη διαχείριση των μεμονωμένων hot spot, αλλά τις δυνατότητες των αρχών να μεταφέρουν ε, τα παιδιά αλλού. Τώρα, κατά πόσο ο διευθυντής ή διοικητής ε, επιβάλλει προστατευτική κυδαιμονία, είναι ένας ε, κίνδυνος που αναλαμβάνουν. Δηλαδή, προτιμούν να μην εξαφανιστούν τα παιδιά. Καλύτερα να έχουν αυτή την ε, προστατευτική κυδαιμονία. Είναι ένα μέτρο εξισορρόπη, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος της εξαφάνισης. Τώρα, ως προς τη διαφυγή, φυσικά τα παιδιά δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις, θέλουν να μετακινηθούν προς άλλα κράτη-μέλη, αλλά αυτό δεν πρέπει να επιληθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και φυσικά, όπως είπατε, αυτό αφορά και τα κριτήρια υποδοχής. Δυστυχώς, η υποδοχή δεν είναι επαρκής για την ευημερία των παιδιών και τουλάχιστον όχι για πολλούς μήνες. Όπως είπατε, ως προς τα κριτήρια υποδοχής, τα πρότυπα υποδοχής θα πρέπει να βελτιωθούν. Αυτά είναι, αυτό είναι ένα από τα βήματα. Και αυτό αφορά και προσωπικό προστασίας των παιδιών που δεν υπάρχει σε πολλά hot spot. Εκτός hot spot τώρα και σε εθνικό επίπεδο και στο μέτρο της δυνατής υποστήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά δεν παραμένουν στα hot spot περισσότερο από όσο χρειάζεται, ιδιαίτερα τα ασυνόδευτα παιδιά, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να βγουν από τα hot spot. Και επίσης, το ανεπαρκές σύστημα μεταφοράς των παιδιών θα πρέπει να βελτιωθεί, έτσι ώστε να μεταφερθούν στη στερεά Ελλάδα ή αλλού θα πρέπει να τύχουν υποστήριξης, να υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες και όχι εις βάρος της ποιότητας ε, της ε, φροντίδας. Μπορεί κανείς να τοποθετήσει σε ένα ε, κτίριο τον διπλάσιο αριθμό παιδιών, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να βλάψει τη φροντίδα και την ευημερία του. Είπατε ότι τα δικαιώματα των παιδιών είναι καθολικά. Είπατε ότι ό,τι συμβαίνει θα πρέπει να ποσοστοποιηθεί και να κρίνουμε και ποιοτικά πόσο ε, είναι για να αντιμετωπιστεί. Ορισμένα ζητήματα είναι πιο επίγοντα, άρα μπορούν να επιληθούν σε επίπεδο hotspot, αλλά όμως όχι. Θα πρέπει να αναλυφθεί ε, δράση σε εθνικό επίπεδο από τις κυβερνήσεις και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει η ιδεώδης λύση, αλλά ως προς τα δικαιώματα των παιδιών, αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα, απόλυτη προτεραιότητα, γιατί βλέπουμε πολύ νέα παιδιά, παιδιά, παιδιά, τα οποία προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, βρίσκονται εκτός, εκτός συστήματος εκπαίδευσης για χρόνια, τέσσερα χρόνια. Και αυτό που βλέπουν στην Ευρώπη δεν είναι αυτό που θα ήθελαν. Και δεν θέλουμε αυτή να είναι η εικόνα της Ευρώπης για το μέλλον, δηλαδή η αντιμετώπιση των παιδιών που προσπαθούν να διαφύγουν από μια εμπόλεμη κατάσταση. Προτρέπουμε λοιπόν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προσπαθήσουν να κάνουν περισσότερα και καλύτερα γνωρίζοντας ότι έχουν αναλυφθεί θετικά μέτρα αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα. Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ και στο δικό σας ερώτημα, αλλά σε αυτά που είπε η κυρία Σίπελ, ξέρετε, ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Φράχη, κάνει πολλά για τα θύματα, με βάση και την Οδηγία Προστασίας των Θυμάτων, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να αποτιμηθεί σε επίπεδο hot spot. Και ειλικρινά, δυστυχώς ε, δεν ε, ακολουθούνται μέχρι τέλους αυτές οι διαδικασίες, γιατί δεν υπάρχουν ε, ε, καταγγελίες, καταγγελίες ε, βιοπραγιών και υπάρχουν και τόσο καυτά ζητήματα που μερικά δεν, μπορούν, δεν μπορούμε να τα δούμε σε επίπεδο hot spot. Πρέπει να βοηθήσουμε τα θύματα, αυτό είναι προτεραιότητα, αλλά η μη κυβερνητική και ε, οι εθελοντές είναι αυτοί που τα αντιμετωπίζουν. Και παρά τις προσπάθειες των εθνικών οργανισμών και φορέων, αυτό είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται κατά προτεραιότητα. Τώρα σε σχέση με την ε, εμπορία και τη, τις βιοπραγίες των διακινητών γνωρίζουμε πολύ καλά αυτές τις καταγγελίες. Δεν τις έχουμε αντιμετωπίσει λεπτομεριακά, γιατί κάτι τέτοιο ε, θα πρέπει να γίνει εκβαθέων. Η κατάσταση είναι τρομακτική, αναμφίβολα. Η καταπολέμηση της ε, εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητες ε, με την επίλυση των άλλων προβλημάτων της μετανάστευσης. Άμεσα στα hot spot δεν ε, υπάρχουν πάντα καταγγελίες, αλλά η Europol καλύτερα πιστεύω ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Η Europol προσπαθεί να προειδοποιήσει και να ειδοποιήσει τις εθνικές αρχές, αλλά το θέμα έγκυται στις εθνικές αρχές να απαντήσουν με σπουδή. Γιατί οι ευάλωτοι άνθρωποι που εντοπίζονται ξαφνικά εξαφανίζονται από τα hot spot. Μιλήσαμε για την περίπτωση Νιγηριανών ε, ε, γυναικών που αποτέλεσαν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, αλλά είναι και οι μόνες. Ακούσαμε και για άλλες παρόμοιες καταστάσεις, αλλά δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Τώρα, σε αυτά που είπε η κυρία Σίπελ, αυτό αφορά την παρουσίαση του συναδέλφου για το Δουβλίνο Μπορώ να πω όμως ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη θεωρούν τις επιστροφές από το Δουβλίνο με βάση τη συνθήκη του Δουβλίνου προς την Ελλάδα ότι αποτελούν ε, αντικείμενο αποφάσεων του ΔΕΚ και θα πρέπει να αποφευχθούν μέχρι ότου αλλάξει η κατάσταση στην Ελλάδα και όταν μειωθεί το άχθος ε, προς την Ελλάδα αυτό το μεγάλο φορτίο της Ελλάδας. Μιλώ από την άποψη της ΦΡΑ, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι η ε, απάντηση στην κυρία Σίπελ αφορά το επόμενο, την επόμενη παρουσίαση. Τελική ερώτηση την κυρία Βίνμπεργκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κατανοώ ότι υπάρχουν πολλά χάσματα σε σχέση με την αντιμετώπιση της κατάσταση ε, ως προς την διέλευση των συνόρων και ε, η διέλευση των συνόρων από Ελλάδα προς Ιταλία δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με τα μία συνόδευτα παιδιά είπατε ότι κάνετε ελέγχου, αλλά δεν είπατε πώς διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι. Βασιζόσαστε στα λεγόμενα αυτών των παιδιών, των ανηλίκων ή δεν ξέρω Πώς κάνετε, τι κάνετε, ακτινογραφίες, πώς κάνουν ε, σε άλλες χώρες. Μας είπατε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί πολλοί ανήλικες δηλώνουν ότι είναι ενήλικες για ευνόητους λόγους. Ε, δηλαδή αυτά τα παιδιά είναι κάτω των 18 και αν το πούν είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφερθούν αλλού στην Ευρώπη θα παραμείνω στην Ελλάδα ή στην Ιταλία. Λένε λοιπόν ότι είναι άνω των 18 γιατί θέλουν να πάνε προς τον Βορρά. Αυτά, αυτά είναι τα δικά μου δεδομένα. Απαντήσεις σε αυτό και σε ακούσουμε μετά την επόμενη παρουσίαση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Πολύ σύντομα να απαντήσω. Καταρχάς, προφανώς δεν είναι ο δικός μας ο οργανισμός ο οποίος κάνει κάποια αξιολόγηση επιτόπου. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται από εθνικές αρχές σε περίπτωση που υπάρχει αφιβολία ως προς την ηλικία του εξεταζόμενου ατόμου. Μιλάμε για κάποιες οριακές περιπτώσεις, εν γέννη και στις δύο χώρες. Δίδεται προτεραιότητα στις δηλώσεις που γίνονται καλή την πίστη από τον ενδιαφερόμενο κάθε φορά. Δηλαδή αποδεχόμαστε ότι αυτός ο οποίος λέει ότι είναι ανήλικος είναι όντως ανήλικος και το αντίστροφο. Γίνονται όμως κιόλας και αξιολόγηση από τις επιτόπου αρχές με διάφορους τρόπους. Μία μέθοδος είναι όντως ο ιατρικός έλεγχος, ένα ιατρικό τσεκάπα. Και όσον αφορά το άλλο τμήμα της ερώτησής σας, όντως στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία, υπάρχει μία γενικότερη τάση ορισμένων ασυνόδευτων παιδιών να λένε τελικά ότι είναι ενήλικες, γιατί πιστεύουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να διαφύγουν πιο εύκολα από τα hot spots. Περισσότερο το βλέπουμε αυτό στην Ιταλία. Στην ε, Ελλάδα υπάρχει ένας γεωγραφικός περιορισμός μετακίνησης, ακριβώς επειδή βρίσκονται πάνω σε νησιά κυρίως αλλά ακόμα και εκεί ορισμένα παιδιά ενδεχομένω να θεωρήσουν ότι είναι καλύτερο να πούν ότι είναι ανήλικε, προκειμένου να καταφέρουν να παραμείνουν στο ανοιχτό τμήμα του hotspot, που θα του επιτρέψει κάποια στιγμή ενδεχομένω να διαφύγουν από το hotspot. Αυτή τη στιγμή γίνει η καταγραφή του. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν πιο εύκολα να μείνουν ενδεχομένω με συγγενεί ή με φίλου, με άτομα με τα οποία έχουν ταξιδέψει και τα οποία ενδεχομένω να βρίσκονται στο ανοιχτό τμήμα του hotspot. Σα ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Ας περάσουμε τώρα στην παρουσίαση του κυρίου Τάμας Μόλναρ. Θα μας παρουσιάσει μια γνωμοδότηση που ζήτησε και πάλι δική μας η Κοινοβουλευτική Επιτροπή όσον αφορά τον αντίκτυπο που θα έχει αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου στα παιδιά. Έχετε το λόγο κύριε Μόλναρ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την πρόσκληση αυτήν, για τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την γνωμοδότηση αυτήν. Κυρίες και κύριοι, εξιότυπα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ σύντομα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα βασικά πορίσματα της γνωμοδότησης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου. Βλέπετε εδώ πέρα στη διαφάνεια κάποια βασικά χαρακτηριστικά του κανονισμού αυτού. Η δική μας η ανάλυση επικεντρώθηκε κυρίως στη νομική πτυχή της αναθεώρησης αυτής. Η γνωμοδότηση λοιπόν διαρθρώνεται σε πέντε σημαντικά σημεία. Θα σας αναλύσω τα σημεία αυτά κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μου. Το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο σημείο το οποίο θίγουμε είναι το ακόλουθο. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, ορισμένοι ετούντες θα αποκλειστούν από το σύστημα του Δουβλίνου. Δηλαδή, θα προβλεφθεί μια νέα διαδικασία επιπαραδεκτού, προτού αρχίσει να ισχύει ο αυτό, αυτός, ένα προκαταρκτικό δηλαδή στάδιο και επομένω θα αποκλείεται η εξέταση ορισμένων ετούντων ετούντες άσυλο, οι οποίοι έρχονται από μία άλλη χώρα, από μία άλλη χώρα πρώτης εισόδου ή από συγκεκριμένε κατηγορίες τρίτων χωρών. Προβλέπεται εδώ πέρα μια ειδική διαδικασία επί του παραδεκτού της αίτησής τους. Οι ειδικέ αυτές διαδικασίες μπορεί ενδεχομένω να επηρεάσουν τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση, την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπω προκύπτουν από τη Σύμβαση των Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Υπάρχει και μια τέταρτη κατηγορία, σε άσυλο εκείνοι, οι οποίοι αποτελούν ή ανταποκρίνονται σε σημαντική απειλή για τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια. Αυτοί θα διοχετεύονται, αν μπορώ να το θέσω έτσι, σε μια προκαταρκτική διαδικασία πάλι προτού αρχίσει να ισχύει ο κανονισμό του Δουβλίνου. Όταν όμω πρόκειται για παιδιά τα οποία ενδεχομένω ανταποκρίνονται σε απειλή, σε κίνδυνο όσον αφορά τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια, συνήθω αναφερόμαστε σε ανήλικους οι οποίοι ανταποκρίνονται σε περίπλοκες περιπτώσεις και οι οποίοι έχουν ειδικέ ανάγκες. Ακριβώς επειδή είναι περίπλοκες όμως περιπτώσεις αυτές, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία τους και θα πρέπει να ακολουθούν εδώ πέρα δίκες διαδικασίες. Αν δεν βρεθεί λοιπόν απαραίτητος αυτός χρόνος για την εξέταση των αιτήσεών τους, τότε αυτό μπορεί να έχει αρνητικέ επιπτώσεις για την προστασία των παιδιών και για την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών, σύμφωνα πάλι με την ε, Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Λέμε εμεί και πάλι ότι τα παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες θα πρέπει να αποκλείονται από το στάδιο αυτό προτού αρχίσει να λειτουργεί η διαδικασία του Δουβλίνου. Όσον αφορά τώρα τις α, παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις, πάλι εδώ πέρα προβλέπεται ένα συγκεκριμένο σύστημα στα πλαίσια του νέου κανονισμού του Δουβλίνου και προβλέπονται εδώ πέρα μια σειρά από κυρώσεις ή ε, μια σειρά από άλλους περιορισμούς που θα μπορούσαν να επιβληθούν στα άτομα αυτά προκειμένου να αποφευθεί η παράτυπη δευτερογενής μετακίνηση. Προβλέπεται λοιπόν ότι ένας ετών θα μπορούσε να προωθηθεί προς την αρχική χώρα εισόδου και θεωρούμε πάντως ότι τα όσα προβλέπονται εδώ πέρα σε σχέση με τα μέτρα τα περιοριστικά μπορεί τελικά να αντιβαίνουν στο μίσον συμφέρον του παιδιού καθώς επίσης και στα δικαιώματα προσφυγής που θα πρέπει να έχει τόσο το παιδί όσο και ένας ενήλικας. Στην γνωμοδότηση λοιπόν λέμε ότι τα μία συνόδευτα παιδιά που αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού θα πρέπει να εξαιρούνται από τις διαδικασίες καταπολέμησης της παράτυπης δευτερογενής, δευτερογενούς μετακίνησης. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί έτσι ώστε να αποκλείονται πάλι τα παιδιά από τις διαδικασίε αυτές, να προβλέπονται συγκεκριμένε προϋποθέσεις προστασίας στην περίπτωση εκείνη που έχουν ήδη υποπέσει σε παράτυπη δευτερογενή μετακίνηση και έχουν ήδη ενταχθεί στη διαδικασία αυτή των κυρώσεων. Πάλι εδώ πέρα υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα συμβατότητας με το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, την ακαιρεότητα και ελοχεύει ο κίνδυνος της μη σωστή μεταχείριση των παιδιών αυτών και τη μη τήρηση των ε, δικαιωμάτων του. Θα πρέπει λοιπόν το παιδί να έχει πρόσβαση επίση στη υγειονομική περίθαλψη, σε εκπαίδευση και αυτό το ζήτημα μπορεί να τεθεί λοιπόν. Και η νομολογία των δύο δικαστηρίων στην Ευρώπη, δηλαδή και το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, περιορίζουν τη δικαιοδοσία των κρατών μελών όσον αφορά τις διαδικασίες αυτές αντιμετώπισης της παράτυπης δευτερογενούς μετακίνησης. Η δική μας λοιπόν γνωμοδότηση λέει ότι θα πρέπει ήδη στην ιδεολογική σκέψη του κανονισμού να φαίνονται ότι υπάρχουν κόκκινε γραμμέ, συγκεκριμένα όρια πέρα από τα οποία δεν μπορούμε να πάμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περίσταση θα τηρούνται τα δικαιώματα του παιδιού. Επίσης προβλέπονται πολλές φορές περιορισμοί στην ε, υποβολή αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό πάλι περιορίζει την τήρηση του μείζωνος συμφέροντος του παιδιού και περιορίζει τη δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης για κάποια παιδιά. Εμείς θεωρούμε ότι οι προθεσμίες οι χρονικές προβλέπονται στην πρόταση κανονισμού θα πρέπει να διαγραφούν και θα πρέπει να, να επιστρέψουμε στο υφιστάμενο καθεστώς που έχουμε στον ισχύοντα κανονισμό. Τέλος, αν η πρώτη αίτηση αποσυρθεί, τότε η δυνατότητα υποβολής μιας δεύτερης αίτησης ασύλου ενδεχομένως να μην χαίρει μιας ουσιαστικής εξέτασης των νέων στοιχείων. Αυτό το οποίο βλέπουμε πολλές φορές είναι όταν έχει υποβληθεί μια πρώτη αίτηση και έχει απορριφθεί και υποβάλλεται στη συνέχεια μια δεύτερη αίτηση η οποία δεν περιλαμβάνει νέα ή σημαντικά νέα πραγματικά περιστατικά, τότε η δεύτερη αυτή αίτηση δεν τυχαίνει τη σωστή μεταχείριση. Είναι σημαντικό λοιπόν εμεί να διασφαλίσουμε, ιδίω όταν πρόκειται για ανήλικου ή για παιδιά, ότι η δεύτερη αυτή αίτηση χορήγηση ασύλου όντω εξετάζεται ολοκληρωτικά, εντελεχώς. Αναφερόμαστε έπειτα στις διασφαλίσεις, τις δικονομικές, τις διαδικαστικές για τα παιδιά. Όντως προβλέπουν εδώ πέρα κάποιες πρόνοιες στον κανονισμό που όντω ενισχύουν την κατάσταση του παιδιού. Λέμε ότι θα πρέπει το παιδί να ενημερώνεται με τρόπο φιλικό προς το παιδί. Όντως η υποχρέωση αυτή δεν υφίστατο στον, στον υφιστάμενο κανονισμό, θα πρέπει να υπάρξει πάντως στον νέο κανονισμό. Επίσης προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις παρεκκλήσεις όσον αφορά τη δικασία διεξαγωγής συνέντευξης και επίσης ότι θα πρέπει να δίδεται τη δυνατότητα στο παιδί να προσφεύγει νομικά και να έχει δικαίωμα σε μία αποτελεσματική δικαστική ακρόαση. Θεωρούμε πάλι εδώ πέρα ότι θα πρέπει να δίδεται τη δυνατότητα για τους ασυνόδευτου ανήλικες και για τα παιδιά να υποβάλουν και νέα στοιχεία ή να συμμετέχουν σε προσωπικες συνεντεύξει και ακροάσεις ακόμα και μετά το τελος της προκαταρκτικης αυτης διαδικασιας που προβλέπεται στον κανονισμό του Δουβλίνου. Αυτή τη στιγμή το σύστημα ως έχει δεν δίνει τη δυνατότητα αυτή και ούτε προβλέπει τη δυνατότητα πρώτερης προσωπικής συνέντευξης. Επίσης, θα πρέπει να δίδεται τη δυνατότητα υποβολής νέων στοιχείων όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση. Πολλές φορές ε, βλέπουμε ότι στο νέο κανονισμό το βάρος των αποδεκτικών στοιχείων τελικά βαρύνει τώρα περισσότερο τον ετούντα. Θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται αποτελεσματικά για την συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, βοηθώντας κατά αυτόν τον τρόπο τον εντούντα άσυλο και αυτός ο επιμερισμένος τρόπος συλλογής αποδεικτικών στοιχείων επιβεβαιώνεται και από την νομολογία των δικαστηρίων, του δικαστηρίου μάλλον του Στρασβούργου. Όσον αφορά τώρα την προστατευτική κυδαιμονία, και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να ισχύει και να μην αποτελεί απλώς μία νομική εκπροσώπηση του παιδιού. Ήδη στη γνωμοδότηση για τα hot spots αναφερθήκαμε τα εθνικά συστήματα κυδαιμονίας. Στη νέα πρόταση λοιπόν του κανονισμού του Δουβλίνου δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο την νομική εκπροσώπηση των παιδιών, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα και τη διατύπωση που χρησιμοποιείται και σε άλλα νομικά μέσα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του ασύλου. Δηλαδή να λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε έναν πραγματικό κυδαιμόνα, ένα άτομο ή μία αρχή που θα μπορούσε πραγματικά να εκπροσωπήσει και να προωθήσει το μείζον συμφέρον του παιδιού. Αυτό λειτουργεί λοιπόν υπέρ προφανώς του συμφέροντος του παιδιού και τηρεί κατά αυτόν τον τρόπο και το το δικαίωμα του παιδιού σε μία αποτελεσματική προσφυγή. Τέλος, οι προθεσμίες έθεσης σε σχέση με μία αρνητική απόφαση. Αυτή τη στιγμή η χρονική προθεσμία είναι 7 ημέρες. Επίσης, οι εφέσεις αυτές είναι πολύ περιορισμένες όσον αφορά την ε, ουσιαστική αξιολόγηση της αναθεώρησης. Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις ε, επί των οποίων μπορεί μια έφεση να θεωρηθεί παραδεκτή. Θεωρούμε εμεί ότι αυτό το πεδίο εφαρμογή θα πρέπει να διευρυνθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή η πολύ περιοριστική προσέγγιση που υπάρχει στον τομέα των εφέσεων τελικά βάλει κατά του συμφέροντος του παιδιού και των δικαιωμάτων των παιδιών. Εμείς θέλουμε πιο ευέλικτα χρονικά περιθώρια, πιο ευέλικτες προθεσμίες και θεωρούμε ότι ε, η οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογή, η οποία είναι ιδιαίτερα περιοριστική αυτή τη στιγμή όσον αφορά τι εφέσεις, θα πρέπει να διευρυνθεί και να αναφέρεται πλέον σε όλα τα δικαιώματα τα οποία αναφέρονται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε τα χρονικά περιθώρια τα οποία προβλέπονται από τις διάφορες χώρες όσον αφορά το ζήτημα της έφεσης για τις μετακινήσεις στα πλαίσια του συστήματος του Δουβλίνου. Βλέπετε ότι σε πάρα πολλά κράτη-μέλη το χρονικό περιθώριο είναι υψηλότερο τελικά από τις 7 ημέρες. Ορισμένες χώρες φτάνει τις 30 ακόμα και τις 60 ημέρες. Τέταρτον τώρα. Μίσον συμφέρον του παιδιού. Στην περίπτωση των ασυνόδευτων παιδιών που δεν έχουν ε, οικογένεια, ή μέλη της οικογένειάς τους σε κανένα κράτος μέλος της περιοχής του Δουβλίνου. Στην περίπτωση λοιπόν αυτό θα πρέπει να εξετάζουμε την αίτησή του σε ένα κράτος μέλος όπου μπορεί να προωθηθεί το μείζον συμφέρον του παιδιού. Εν προκειμένου, δεν αναφερόμαστε στο κράτος μέλος της πρώτης νόμιμης εισόδου ή στο κράτος μέλος εκείνο το οποίο έχει θεωρηθεί υπεύθυνο με βάση τους γενικούς κανόνες προκειμένου να εξεταστεί σε πρώτη φάση το συμφέρον του παιδιού. Θα πρέπει να τροποποιηθεί με άλλα λόγια η πρόταση αυτή με βάση την υφιστάμενη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπονται οι κατάλληλες διαδικασίες για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου Λέμε λοιπόν εμείς ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πολύ ε, τομεακή πολυεπιστημονική ομάδα με τη συνεργασία του και του παιδιού κατά την αξιολόγηση των, ε, του μείζοντος συμφέροντος του παιδιού. Κατά αυτόν τον τρόπο η διαδικασία θα καταστεί πολύ πιο αποτελεσματική. Τώρα θα πρέπει να έχουμε το σωστό μηχανισμό κατανομής όσον αφορά τα παιδιά η δυνατότητα της οικογενειακής επανένωσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι το πρώτο κριτήριο. Σε περίπτωση δηλαδή μετακίνηση του παιδιού σε κάποια άλλη χώρα, σε παιδί, περίπτωση μεταγκατάστασης, θα πρέπει το πρώτο κριτήριο να είναι η οικογενειακή επανένωση. Προκειμένου αυτό να λειτουργήσει αποτελεσματικά θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο να ενσωματωθεί στην νομοθετική αυτή πράξη. Έπειτα, την τελική ευθύνη για την μετεγκατάσταση θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αρχές. Η απόφαση αυτή μπορεί βέβαια να επηρεάσει τα δικαιώματα του παιδιού. Προκειμένου λοιπόν η απόφαση αυτή να είναι συμβατή με τα δικαιώματα του παιδιού, θα πρέπει οι νέες αυτές πληροφορίες για τα μέλη της οικογένειας να επιτρέπονται. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να τροποποιηθεί το κείμενο του κανονισμού προκειμένου να υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις βάσει των οποίων μπορούν να επανανοθούν κάποιες οικογένειες. Δεν θα πρέπει να αποκλείεται οποιαδήποτε παρέκκληση όπως φαίνεται ότι υφίσταται αυτή τη στιγμή ως κανονισμός. Έπειτα, η πρόταση αυτή αναθεωμένη, λέει, αναθεωρημένη, με λέει ότι θα πρέπει συγκεκριμένοι μόνο λόγοι οικογενειακής επανένωσης να δώσουν το δικαίωμα για νέα αίτηση ή να δίνει το δικαίωμα σε κάποιες συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες των παιδιών. Παιδιά, για παράδειγμα, τα οποία έχουν ε, υποστεί ψυχολογικά τραύματα. Θεωρούμε εμεί ότι ε, αυτή τη στιγμή το πεδίο εφαρμογή όσον αφορά τι ανθρωπιστικέ ρήτρε θα πρέπει να διατηρηθεί, να μην περιοριστεί, να καλύπτονται λοιπόν όλες οι ευάλωτε ομάδες. Έπειτα, ο μηχανισμός κατανομής. Καταρχάς, θα πρέπει πάλι εδώ πέρα να δούμε τι ακριβώς προβλέπετε όσον αφορά την συμβολή των εισαγγελέων. Αν οι δημόσιες αρχές στις ε, χώρες ε, προέλευσης έχουν στοιχεία όσον αφορά την οικογενειακή πανένωση, προφανώς μπορούν να συμβάλλουν. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και ένα σύστημα σαν το Eurodac, στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες. Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων των παιδιών, που αυτή τη στιγμή είναι 10 χρόνια, δημιουργεί κάποια προβλήματα συμβατότητας με τα δικαιώματα του παιδιού και με την ε, αρχή του περιορισμού της ε, διατήρησης των δεδομένων αυτών. Θεωρούμε λοιπόν ότι η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα ε, μακροχρόνια, δεν προβλέπεται καμία ευελιξία. Αυτό προφανώς θα πρέπει να τροποποιηθεί. Οι προειδοποίησεις, οι καταχωρήσει προθοποιήσεων που γίνονται σε σχέση με τα παιδιά και αυτό το σύστημα θα πρέπει να τροποποιηθεί. Τα κράτη-μέλη θα, θα πρέπει να μπορούν να απορρίπτουν κάποιες αιτήσει βάσει των απειλών εθνικής ασφάλειας. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι η απόρριψη μιας αίτησης αυτής δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος των δικαιωμάτων του παιδιού και σε καμία περίπτωση θα πρέπει να εισάγει διακριτική μεταχείριση. Προκειμένου λοιπόν το σύστημα αυτό απόρριψη αιτήσεων ασύλου να συνάδει με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα πρέπει για κάθε απόρριψη να υπάρχει μία εξατομικευμένη αιτιολόγηση με καταγραφή όλων των λόγων. Έπειτα, η πιο στενή έννοια τη οικογένεια για τον διορθωτικό μηχανισμό έχει επιπτώσει σε διάφορα άρθρα για τα δικαιώματα του παιδιού. Ο μηχανισμός αυτός κατανομής για τις οικογένειες προβλέπεται τώρα στο γενικό ορισμό του κανονισμού. Εμείς στη γνωμοδότησή μας λέμε ότι όχι μόνο η άμεση οικογένεια, αλλά και οι συγγενείς, οι συγγενείς θα πρέπει να καλύπτονται στην έννοια της οικογένειας. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να προβλεφθούν κάποιες νέες διατάξεις όσον αφορά τον ορισμό της ε, οικογένειας. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδελεχή αυτή ανάλυση. Κύριε Βίξτρομ, θα σας δώσω προφανώς το λόγο. Ήθελα απλώς να πω ότι ε, η παρουσίαση αυτή είναι σίγουρα πάρα πολύ χρήσιμη, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για την εισηγήτριά μας την κυρία Βίξτρομ γιατί πραγματικά μας κάνατε μια πολύ λεπτομεριακή ανάλυση των επιπτώσεων του νέου αυτού κανονισμού και είμαι σίγουρος ότι η παρουσίαση αυτή θα τροφοδοτήσει την, πολλές ερωτήσεις, καθώς επίσης και την ίδια την εισήγηση της κυρίας Βίκστρομ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εντυπωσιακή ε, μελέτη. Με κάνει να αισθάνομαι ότι επιτέλους μπορώ να ανασάνω πιο ελεύθερα, γιατί συμμεριζόμαστε κοινέ απόψεις ως προς τη διαδικασία εισδοχής, αλλά οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σημαίνει, σημαίνουν ότι θα πρέπει να συλλεγούν στοιχεία για τα μέλη της οικογένειας. Εσείς αναφέρεστε στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά για ποιες υποθέσεις, σε ποιες υποθέσεις. Επίσης, επ' αυτού του θέματος ως προς την κυδαιμονία στην οποία αναφερθήκατε. Εμείς χρειαζόμαστε όχι μόνο μια πλήρη κυδαιμονία, αλλά ένα σύστημα προστασίας για τα παιδιά. Και η ομάδα που προτείνεται είναι μία από τις ιδέες αυτές, αλλά απέχει πόρο από την πραγματικότητα για την οποία άκουσα σήμερα. Μου δώσαν ορισμένα αριθμητικά στοιχεία ε, και μου ελέγχθη ότι στην Ιταλία ότι ένας μπορεί να έχει την κυδαιμονία 300 ατόμων. Αυτό δεν είναι αποδεκτό γιατί είναι εύκολος ο διορισμός, αλλά αν κάποιος είναι κηδεμόδας εκατοντάδων ή χιλιάδων ασυνόδευτων παιδιών, τότε η έννοια της κυδεμονίας έχει χάσει τη σημασία της. Χρειαζόμαστε ένα πακέτο, μία προσέγγιση πακέτου, όπου λαμβάνεται υπόψη και η κυδαιμονία και όπου χρειάζονται επαρκείς πληροφορίες σε μία γλώσσα που είναι κατανοητή από τον ενδιαφερόμενο με νομικές συμβουλές και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα επιλύονται ως διαμαγείας με το διορισμό κηδεμόνα. Το είδατε αυτό. Θα μπορούσαμε να το συζητάμε επί Α, και κάτι άλλο. Ως προς τις ε, προθεσμίες, την προθεσμία έφεσης ε, που είναι 7 ημέρες, εσείς είπατε ότι θα πρέπει να είναι ευέλικτη και ότι θα πρέπει το πεδίο εφαρμογής να μην ισχύει. Τι εννοείτε με αυτή την ευελιξία. Θα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θα επανέλθω ε, σε λίγο αν οι συνάδελφοι δεν θίξουν άλλα ερωτήματα. Σεσίλια, θέλω να ρωτήσω κατά πόσο υπάρχουν ε, ερωτήσεις. Μπίργκιτ, ε, ε, κάτι σύντομο, μια σύντομη παρέμβαση, γιατί τα καταφέραμε πολύ καλά χρονικά, αλλά δεν πρέπει να υπερβούμε τα χρονικά μας όρια. Θα ε, επανέλθω στο θέμα επιστροφής των ενδιαφέρομενων και ξέρω ότι αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό του Δουβλίνου μπορεί να γίνει επιστροφή προσφύγων, αλλά αναφέρθηκα και στη ΦΡΑ, γιατί πολλά κράτη-μέλη δεν ε, προσφεύγουν σε αυτή λόγω κατάστασης και ο οργανισμός, η ΦΡΑ λέει ότι χαίρεται γιατί επί του παρόντος τα κράτη-μέλη δεν το κάνουν. Δέχομαι αυτή την ιδέα και θα ήθελα να δηλώσω ότι δεν χαίρομαι γιατί η Επιτροπή ε, μιλά για ένα συμβουλευτικό πλαίσιο για την επιστροφή προσφύγων στην Ελλάδα. Και εδώ μιλάμε για παιδιά και ενηλίκους. Επίσης έχω και ένα ε, ερώτημα ως προς το εξής τι πιστεύετε ως προς το μελλοντικό, ένα μελλοντικό σύστημα του Δουβλίνου. Δηλαδή όταν η επιστροφή προσφύγων είναι υποχρεωτική και όχι ένα από τα ενδεχόμενα όπως ε, συζητείτε. Ως προς το μη παραδεκτό, τη μη παραδοχή, εδώ δεν μιλάμε μόνο για το ότι η οικογενειακή επανένωση δεν τηρείται. Είπατε ε, για την ε, ε, έλευση στην πρώτη χώρα, προέλευση από τρίτες χώρες και ούτω καθεξής. Και φυσικά δεν μπορούμε να αναλάβουμε όλους τους πρόσφυγες, αλλά με όλους αυτούς τους κανόνες δημιουργούμε την εντύπωση ότι στο τέλος δεν θέλουμε να αναλάβουμε κανέναν. Γιατί έχουμε τη, την Τουρκία, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες που δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλείς. Μπορείτε να μας πείτε πώς το βλέπετε και πείτε μου αν σφάλω. Ευχαριστώ, Μπίργκιτ. Η κυρία Σέμενεκ παρακαλώ να είναι ιδιαίτερα σύντομη. Ο κύριος Σέμενεκ. Ε, ε, δεν θα ήθελα να σχολιάσω τη δήλωση της Μπρατισλάβα. Είναι κάτι το οποίο έχει εγκριθεί εκτός ε, της επιρροής του Συμβουλίου και εκτός Προεδρίας. Το ζήτημα είναι κατά πόσο προσδίδει σημασία η Προεδρία στην κατάσταση των ανηλίκων. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι το κάνει και ε, ίσως θα χαρείτε να μάθετε ότι το δεύτερο ημισή του Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με συλλογή στοιχείων με βάση το IPCR, δηλαδή την ε, ολοκληρωμένη κατάσταση ε, αποτίμησης για τους ε, ανηλίκους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Φρά για το input που μας έδωσε. Πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για την εξαφάνιση ανηλίκων ή εκείνους που ε, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης ή εγκληματικών ενεργειών. Η Προεδρία προσδίδει μεγάλη σημασία σε αυτά. Ε, ζητώ συγγνώμη κύριε Σέμενεκ που σας είπα να είσαστε σύντομος, αλλά δεν έχουμε χρόνο. θα ζητήσω αν γίνεται να απαντήσετε σε σχέση και με αυτά τα θέματα αυτά. Πέντε λεπτά για να μπορέσετε να τοποθετηθείτε. Χρειάζεστε σαφώς περισσότερο χρόνο, αλλά πρέπει να περιοριστούμε. Θα ήμουν ευγνώμων. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Με πέντε λεπτά να μπορέσετε να τοποθετηθείτε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε πέντε λεπτά να συμπιέσω τις απαντήσεις μου. Πρώτον, όσον αφορά τον επιμερισμό υποχρεώσεων, όσον αφορά τα κράτη-μέλη, η αναφορά σε σχέση με την ομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια υπόθεση του 2012 δηλαδή σε σχέση με τα δικαστικά θέματα και την, την Ιρλανδία. Είναι δηλαδή η συγκεκριμένη αυτή η περίπτωση που θέτει αυτή την υποχρέωση. Συμφωνώ απόλυτα με την ανάγκη σας να υπάρχει ένα βελτιωμένο πλαίσιο και με ένα καλύτερο πλαίσιο κυδεμονίας να μπορέσουμε να ε, δράσουμε. Είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε και από πλευράς ε, ε, συναδέλφων όσον αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με τα όσα ζητείτε να γίνουν και σε σχέση με τις δράσεις όσον αφορά την πρόταση αυτή από πλευράς διατάξεων και προδιαγραφών τι θα έπρεπε να γίνει όχι μόνο σε σχέση με το σχεδιασμό αλλά και με τη δράση επιτόπου όσον αφορά την ερώτηση προθεσμιών, διοριών και πώς αυτό θα μπορούσε σε ένα ευέλικτο πλαίσιο να δράσει. Έχετε δίκιο σε αυτό. Σε άλλα μέσα ο το εύλογο διάστημα είναι μια έννοια που αναπτύσσεται από πλευράς νομολογίας της ε, Ένωσης. Κάτι δηλαδή γύρω από αυτό το εύλογο πρέπει να υφίσταται, δίνοντας ένα περιθώριο δράσης για τα κράτη-μέλη, αλλά επίσης ε, και αναγνωρίζοντας τα κριτήρια, τα, τους περιορισμούς όσον αφορά τα κριτήρια που περαιτέρω όσον αφορά την ανάπτυξή τους από πλευράς νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευελιξία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά σε σχέση με τις ερωτήσεις της κυρίας Τσίπερ. Ο έλεγχος αποδεκτού, παραδεκτού θέτει και ζητήματα φυσικά ταυτοποίησης. Όμως ε, αυτό το οποίο υπάρχει ως ε, θέμα, το οποίο υφίσταται ως στις διαδικασίες και προδουβλίνου, είναι να βασίζεται κανείς στην έννοια των ασφαλών χωρών, ασφαλών τρίτων χωρών στην οποία πρέπει να μπορεί να βασίζεται κανείς. Και αυτό έχει και επιπτώσεις όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου και σε σχέση με την αιτιολογημένη γνώμη όσον αφορά την προσέγγιση ασφαλών χωρών Υπό το ίδιο πρίσμα αντιμετωπίζουμε και εμείς αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν ε, δεδομένα σχετικά για να απαντήσω. Βρίσκεται στο πλαίσιο των ε, δυνατοτήτων της υπηρεσίας μας. Δεν θέλαμε εδώ να υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα όσον αφορά τις ασφαλείς τρίτες χώρες. Ωστόσο η γνωμοδότησή μας, η άποψή μας σχετικά είναι ότι αυτή την έννοια, αυτή η έννοια δεν είναι κάτι το οποίο ε, ε, δεν θα μπορούσαμε να ε, λειτουργήσουμε χωρίς αυτό. Ευχαριστώ. Είναι τόσο περίπλοκα τα θέματα και ευχαριστώ για την ε, ε, τοποθέτησή σας όσον αφορά την, τοποθε... την συνθήκη του Δουβλίνου. Να επαναλάβω, θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την υψηλή ποιότητα των παρεμβάσεών σας και για την δική σας προσπάθεια. Ευχαριστούμε για το έργο που επιτελείτε είναι σημαντικό σε σχέση με ένα κείμενο που θα μπορεί να είναι ε, ως βάση για τις δράσεις μας. Θέλω να ευχαριστήσω <clears throat> για την παρουσία και την προσπάθειά σας για αυτή την σημαντική γνωμοδότηση και για την συνεχόμενη αυτή η συνεισφορά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που προσήλθατε. Ευχαριστώ και πάλι. Συνάδελφοι, θα ψηφίσουμε ακριβώς στις 11 η ώρα. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.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 Colleagues, please take your seats. We can begin. Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι να ξεκινήσουμε. I will now do so. Uh, αγαπητοί συναδελφέ, περάσουμε στο σημείο 7 τη σας διάταξη, Οργανισμό Ευρωπαϊκή Ένωση για το Άσυλο. Ψηφίζουμε για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων και για την ομάδα διαπραγματευτών. Ωραία, βλέπω ότι με προσέχετε τώρα. Σήμερα το πρωί, αγαπητοί συνάδελφοι, θα κρατήσει η ψηφοφορία περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο, αλλά ενδεχομένως να καταφέρουμε να προχωρήσουμε και πιο γρήγορα. Έχετε τις κάρτες ψηφοφορίας μαζί σας, αν όχι πείτε το μου τώρα. Λοιπόν, έχετε όλες τις κάρτες σας, πολύ ωραία. Ξεκινάμε με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Δύο σύντομες ανακοινώσεις θα ήθελα να κάνω και απευθύνομαι και στον κύριο Νίντερ Μιλέρ. Η κυρία Ματέρα έχει αποσύρει την ε, τροπολογία της, ε, μάλλον την υπογραφή της για την τροπολογία 572. Η κυρία Βόζεμπερκ υποστηρίζει τις ακόλουθες τροπολογίες 239, 261, 274, 355, 307, 426, 338, 343, 344, 366, 380, 383, 490, 393, 504, 522, 528, 529, 578, 599, 642, 645, 653, 654, 677 και 684. Δεν ξέρω αν ο συγητής ο κύριος Νίντερ θέλει να πάρει τώρα το λόγο πρωτού ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω, πραγματικά να ευχαριστήσω τους γιώδης εισηγητές συναδέλφους διότι υπήρχε πολύ επικοδομητική θετική ατμόσφαιρα επεξεργαζόμενη στην την έκθεση. Ήταν χαρά να συνεργαστώ με τους συναδέλφους αυτούς. Ταυτόχρονα όμως, από την άλλη πλευρά, πρέπει να ευχαριστήσω και τους βοηθούς μου και τη γραμματεία, διότι πραγματικά έκαναν εκείνη την δύσκολη και εξαιρετική αυτή δουλειά. Σας ευχαριστώ όλους σας, εσάς. Μια τεχνικού χαρακτήρα παρατήρηση, μια τεχνική προσαρμογή στον συμβιβασμό 26 επί του άρθρου 35 που σε σχέση με τους σκιώδεις είχε συμφωνηθεί αλλά εκ παραδρομής ε, δεν αναφερόταν στην παράγραφο 4 λοιπόν στο άρθρο 35 η τελευταία πρόταση θα πρέπει να διαγραφεί για να κατανοηθεί καλύτερα αυτό έχουμε το, την εξής, ε, το εξής πλαίσιο η υπηρεσία στο πλαίσιο της συμφωνίας σε σχέση με τρίτες χώρες και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συντονίζει τέτοιου είδους ανταλλαγές πληροφοριών ή άλλου είδους δράσεις σε σχέση με τρίτες χώρες μέσα στο θέμα των επικρατιών αυτών των χωρών. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο επιλύεται το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πέτα Νίντερ Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ψηφίζουμε. Ξεκινάμε. Απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τροπολογία 103. Άρχεται η ψήφιση ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 106 και 128 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. Περνάμε στα άρθρα. Συμβασμός 1 στο άρθρο 1. Παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περνάμε στο συμβιβασμό 1α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Συμβιβασμός 1α. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 2. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Συμβασμός 3. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαθμός 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 5. Άρχεται. Πέρας. εγκρίθηκε. Συμβασμός 6 άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. Συμβασμός 7 άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. Τροπολογία 354 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβασμός 8 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 9 άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. Συμβασμός 10 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Πάμε στο συμβασμό 12, 13 και πρώτο του 15. Άρχεται. Πέρας. εγκρίθηκαν. Δεύτερο τμήμα του Συμβασμού 15 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα του 15 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 14. Άρχεται. Just keep turning your pages. Compromise 14. Just Γυρίστε τις σελίδες σας και το βρείτε. Δεν έχουμε αριθμού σελίδων. Συμβιβασμός 14 λοιπόν. Το βρήκατε. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 16. Άρχεται. πέρας εγκρίθηκε. Τροπολογία 508 άρχεται. 508 παρακαλώ άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. λυπούμε γι' αυτό. Συμβασμό 17 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 18 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 19 άρχεται. πέρας εγκρίθηκε. Συμβασμός 20 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 21 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 22 άρχεται. πέρας εγκρίθηκε συμβασμός 23α άρχεται πέρας εγκρίθηκε συμβιβασμός 23 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 23α άρχεται Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 71. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 72. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε.

απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 23 Β. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 24 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 25 άρχεται. πέρας εγκρίθηκε σύμφωνος 26 άρχεται πέρας εγκρίθηκε σύμφωνος 27 άρχεται εγκρίθηκε Σύμβασμος 28 άρχεται πέρας εγκρίθηκε συμβασμός 29 άρχεται πέρας εγκρίθηκε συμβασμός 30 άρχεται πέρας εγκρίθηκε συμβασμός 31 άρχεται Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 32. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 33. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 35. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 34. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 36. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 37. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 670. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 671. Άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. Σύμφασμος 38 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 39 συμβιβασμός άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 40 άρχεται. Πέρας. εγκρίθηκε. Τροπολογία 675 άρχεται. Δεν μπορούσε να έχει αγνοηθεί να μη συμμετείχαμε. Εντάξει, να δούμε ποια θα είναι η έκβαση. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Δυστυχώς απορρίφθηκε, δυστυχώς λυπούμε. Συμβασμός 41, άρχεται. Ναι, Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το συμβασμό 41. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβασμό 42. Άρχεται. Πέρας. Όχι, δεν θα καταψηφίσετε. Τροπολογία 678. Εγκρίθηκε ο συμβιβασμός. 678 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 43 άρχεται. Πέρας. εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 44 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 683 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Συνάδελφοι, 104 τροπολογία άρχεται πέρας απορρίφθηκε 105 άρχεται πέρας απορρίφθηκε 109 τροπολογία άρχεται πέρας απορρίφθηκε 107 άρχεται πέρας απορρίφθηκε 108 άρχεται πέρας απορρίφθηκε 110 άρχεται πέρας γιατί συνάδελφοι τεχνικό σφάλμα έγινε στην 110. Πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία στην 110 για την αιτιολογική αυτή σκέψη. Ψηφίζουμε λοιπόν. 110 επαναλαμβάνουμε. Άρχεται η ψηφοφορία πάλι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 111 τροπολογία άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβιβασμό 45. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 116 τροπολογία. Άρχεται. εγκρίθηκε 117 άρχεται πέρας απορρίφθηκε συμβασμός 46 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 47 συμβιβαστική άρχεται Πέρας. Εγκρίθηκε. 48. Συμβαστική τροπολογία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 131 τροπολογία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβασμό 49. Άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. Συμβασμός 50 άρχεται. πέρας. Εγκρίθηκε. 51 συμβαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 52 άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. Συμβασμός 53 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 54 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 55 συμβασμός άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. 56 συμβαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 167 άρχεται. 167 πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 58 άρχεται. Πέρας. αιτιολογική σκέψη <clears throat> τροπολογία 3 στο αιτιολογικό άρχεται πέρας εγκρίθηκε 178 τροπολογία άρχεται πέρας εγκρίθηκε 179 άρχεται πέρας απορρίφθηκε 180 άρχεται πέρας απορρίφθηκε 181 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 182 άρχεται πέρας απορρίφθηκε. Συμβασμός 59 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 189 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. 193 άρχεται. Πέρας. εγκρίθηκε 192 άρχεται α συγγνώμη 195 ναι. άρχεται 195 παρακαλώ άρχεται συγγνώμη συνάδελφοι 194 όχι 195 194 άρχεται πολύ μεγάλη αλλαγή. 194 Ψήφισετε όλοι πέρας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 195 τώρα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. 196 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Σύμβασμος 60 άρχεται πέρας εγκρίθηκε συμβασμός 61 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 62 άρχεται πέρας εγκρίθηκε συμβασμός 63 άρχεται Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 64. Άρχεται. Την 64. Δεν την είπα. Συμβαβός 64. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 65. Άρχεται. Πέρας. εγκρίθηκε σύμφασμος 66 άρχεται πέρας εγκρίθηκε σύμφασμος 67 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 218 τροπολογία άρχεται και οι 219 ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκαν. Με συγχωρείτε, απορρίφθηκα 220 τροπολογία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. 221 άρχεται. Πέρας απορρίφθηκε 222 άρχεται πέρας απορρίφθηκε συμβασμός 68 άρχεται πέρας εγκρίθηκε τροπολογία 8 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 9 άρχεται πέρας εγκρίθηκε συμβασμός 69 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 228 τροπολογία άρχεται πέρας απορρίφθηκε 229 άρχεται πέρας απορρίφθηκε 230 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 231 άρχεται πέρας Απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 70. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στα εδάφια, στο 15 του προϋπολογισμού νομοδότησης άρχεται εδάφιο 15 της νομοδότησης για τον τροπολογία 15 παρακαλώ ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας έχετε το σωστό φύλλο τη σωστή τροπολογία είσαστε στη σωστή θέση έχουμε το 15 του προϋπολογισμού πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε και πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις ε, για, από πλευράς προϋπολογισμού το 3 άρχεται αιτιολογική σκέψη 3 άρχεται πέρας εγκρίνεται Ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 36 υπέρ 9 εναντίον 6 αποχές. Και τώρα θα ασχοληθούμε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία και άρχεται η ψηφοφορία. The vote Πέρας. Εγκρίνεται 46 υπέρ 4 κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια. Ξέρω ότι είναι επίπονο, συνάδελφοι, τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά χρονικά. Περνάμε απευθείας στην επόμενη ψηφοφορία για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Μπόνι θέλει να λάβει το λόγο. Α, δεν είναι εδώ. Α, με συγχωρείτε, ο κύριος Μπόνι δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ σήμερα. Άρα ψηφίζουμε απευθείας. Συμβιβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Είσαστε όλοι έτοιμοι. Συμβιβαστική 1. Πέρας. That is Εγκρίνεται. Τέσσερα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται.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 Με συγχωρείτε συνάδελφοι, τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Δώδεκα. Ψηφίζουμε για την 12. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Πρώτο τμήμα, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 26, Αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 22. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα ε, ψηφίζουμε το κείμενο στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 48 υπέρ, 1 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Πόνη. Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε διάλειμμα. Συνεχίζουμε. Όχι, αστειευόμουν, αστειευόμουν. αστειευόμουν. Ε, βρετανικό χιούμορ. Κάκιστο. Uh, να σας πληροφορήσω πριν αρχίσουμε με την ψηφορία της έκθεσης Βερσιά, να σας επισύρω την προσοχή στους συμβασμούς 3, 8 και 13. Στην έκθεση Βερσιά ζητήθηκε ξεχωριστή ψηφοφορία 3, 8 και 13. Αν και δεν φαίνεται στον καταλογό σας, απλώς να το δουν οι συντονιστές τα σημεία 2 και 3, των 8 και 13, των 2 και 8 και το δεύτερο τμήμα του 13 θα εκπέσει εάν περάσει το πρώτο. Εντάξει, είναι σαφές. Είναι σαφές για τους συντονιστές. Μόνικα, Μπίργκιτ και οι υπόλοιποι κυρία Στίβενς. Εντάξει, εντάξει, ωραία. Αρχίζουμε λοιπόν. Συμβιβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. θα μπορούσε να το πει και ο αντιπρόεδρος, έτσι και αλλιώς. Εντάξει, ε, συμβαστική 4, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. 24. τέσσερα, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική θερία, Άρχεται η ψηφοφορία. Α, με συγχωρείτε. Τμήμα 1. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροποδολογία 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 54. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τμήμα 1. Πρώτο τμήμα παρακαλώ, τις 8. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83. 83. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 84. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 85. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 103, άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 105. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 111. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 118 άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 120 άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 122. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 131. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 132, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 133, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Πρώτο τμήμα, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 141, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 142, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 143, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στις ιτολογικές σκέψεις. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 26 υπέρ, 22 κατά, καμία αποχή. Να χαρώ την κυρία Βεργιά και δεν τη ρώτησα βέβαια νωρίτερα αν ήθελε να πάρει το λόγο πριν την ψηφοφορία. Αν έχετε να πείτε κάτι τώρα κυρία Βαζιά. έχετε το λόγο παρακαλώ. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόθερμα όλους τους σκιώδεις συγητές, γιατί καταφέραμε να εργαστούμε πολύ επικοδομητικά, ακόμα και αν το έργο μας ήταν δύσκολο. Καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες πάντως από όλους μας, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα κείμενο αποδεκτό από την πλειοψηφία των συναδέλφων. Λυπάμαι λίγο την τελική ψηφοφορία. Καταλαβαίνω βέβαια πώ ψηφίστε σε ορισμένα σημεία. Να ευχαριστήσω ολόθερμα όλου του συνεργάτε και του κοιόδη ηγητέ. Σα ευχαριστούμε κυρία Βεαζιά, λέει ο πρόεδρο. Συγγνώμη που δεν σα έδωσα το λόγο στην αρχή τη ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, α περάσουμε τώρα στην τελική ψηφοφορία για σήμερα. Τελική λοιπόν ψηφοφορία. Ξέρετε ότι στις 29 Νοεμβρίου αλλά και χθες Δύο τριμερείς διάλογοι λάβανε χώρα όσον αφορά το, την αναθεώρηση του μηχανισμού αναστολής με επιτυχία. Ο κύριος Διάς Δεμέρα είναι ο εισηγητής. Νωρίτερα σήμερα μας παρουσίασε την εξαιρετική του έκθεση. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να το συγχαρώ, καθώς επίσης και όλους και οδησηγητές που εργάστηκαν για την έκθεση αυτή. Κύριε Ντιές Ντεμέρα, θέλετε να πάρετε πάλι τώρα το λόγο ψηφίσουμε όχι. Πάντως ξέρω ότι πήρατε το λόγο νωρίτερα. Συγχαρητήρια λοιπόν άλλη μια φορά και σε εσά και σε όλους και οδησηγητές και σε όλους όσοι εργάστηκαν για το δύσκολο αυτό νομοθέτημα. Προχωρούμε λοιπόν στο κείμενο όπως τροποποιήθηκε μέσω των τριμερών διαλόγων, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Και γκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο η διαδικασία της ψηφορίας και ολοκληρώνεται και η πρωνή μας συνεδρίαση. Η ε, Επιτροπή θα συνεδριάσει και το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.